Well, ladies and gentlemen, it is a pleasure. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά αρχίζουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο σημερίσιας διάταξης είναι η έγκριση αυτής. Ελπίζω να γνωρίζετε ότι το πρώτο θέμα είναι το Διαστημικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Οργανισμός Διαστημικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης το επόμενο σημείο είναι ένας κανονισμός του Συμβουλίου για τον πυρηνικό παροπλισμό και το πρόγραμμα ενίσχυσης της, ε, του του πυρηνικού σταθμού Ιγναλίνα στη Λιθουανία ε, και την ανάκληση του κανονισμού 1369 του 2013. Επίσης, ε, συνεχίζουμε με το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη όσον αφορά την έρευνα ε, και μάλλον την αριστεία στην έρευνα και στην καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε κανένα σχόλιο? Αν όχι, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Όσον αφορά την έγκριση των πρακτικών της 13ης ε, Σεπτεμβρίου, υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά αυτά. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, ε, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας, που είναι η θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα. Η συγκητής μας είναι ο Μασιμιλιάνο Σαλίνη. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. πρόκειται για ένα θέμα στρατηγική σημασία ε, και είμαι πεπισμένο γι' αυτό. Ε, και <clears throat> μάλιστα έχω και διάφορες παρεμβάσεις ε, επί των οποίων επί των οποίων εργάζομαι αφορούν 150 τροπολογίες. Λαμβάνω υπόψη μου το γεγονός ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη σύγκληση πάνω σε μια θέση η οποία μπορεί να ε, γίνει δεκτή κυρίως όσον αφορά αυτό το θέμα το πιο αμφιλεγόμενο ας πούμε αυτό που είναι πιο επικίνδυνο εν πάση περιπτώσει αυτό της διακυβέρνησης δηλαδή όπου ας πούμε για παράδειγμα έχουμε λάβει 100 τροπολογίες που αφορούν ακριβώς και μόνο το θέμα αυτό. όσον αφορά την προσπάθεια εξέβρεσης συμβιβαστικών λύσεων που να συμμερίζονται όσο γίνεται περισσότεροι. Το θέμα της διακυβέρνησης είναι πολύ σημαντικό και μπορώ να δεχτώ τα αιτήματα που προκύπτουν από την πρόταση της Κομισιόν να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια στον καταμερισμό ανάμεσα στην Κομισιόν, στη GSA που θα γίνει πλέον ε, η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για, την, ε, για το διαστημικό πρόγραμμα και την ΕΣΑ. Και λέμε ότι εάν ε, η νέα υπηρεσία GSA, η νέα υπηρεσία δηλαδή για το διάστημα, ε, αν έχει συγκεκριμένες ε, δραστηριότητες και ευθύνες, τα μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Επίσης υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν το downstream και που τα συμμερίζονται και οι ε, σκιώδεις Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και κάποια ε, ιστορικά ε, ισχυρή ικανότητα upstream και λόγω του Γαλιλαίου. Θα πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτό το τμήμα που ορίζουμε ως downstream έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η ε, ε, βιομηχανία μας θα μπορέσει να, να χρησιμοποιήσει συγγνώμη, τις υποδομές που θα έχουμε δημιουργήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρασμα για την ε, υπηρεσία GSA. Απ' την άλλη πλευρά και η ΕΣΑ είναι σημαντικό να ενδυναμωθεί και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τον τεχνικό πυλώνα της ευρωπαϊκής διαστημικής ε, πολιτικής. Αλλά βεβαίως ε, βάσει της διακυβέρνησης ε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την συνεργασία μεταξύ GSA και ESA. Η GSA είναι ενωσιακή υπηρεσία ενώ στην ΕΣΑ συμμετέχουν αρκετές αλλά όχι όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες τρίτες χώρες. Επομένως θα πρέπει να ξεκαθαριστούν νομικά αυτά τα στοιχεία. Να πω και δύο λόγια όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Τα ε, κονδύλια για το διαστημικό πρόγραμμα είναι ικανοποιητικά. Έχουμε 16 δις πρόταση της Κομισιόν, αυτό είναι εξαιρετικό νέο σε σχέση με το παρελθόν. Και στην διατύπωση τροπολογιών, εγώ προσωπικά υποστηρίζω ότι ε, πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε γιατί μιλάμε, να το ξεκαθαρίσουμε με τους, συναδέλφους σχετικά με τα νέα προγράμματα τα οποία είχαν πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση. 500 εκατομμύρια δόθηκαν για το GovSatcom και το ε, ε, SSA με τρόπον ώστε στη συζήτηση με, τη, με τους συναδέλφους ορισμένοι υποστήριξαν και υπογράμμισαν ότι εάν ο προϋπολογισμός είναι τόσο τόσο περιορισμένος, με 250 δηλαδή εκατομμύρια ένα πρόγραμμα, θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να περικοπούν δραστηριότητες. Επομένως, γίνεται μία προσπάθεια να δοθούν επιπλέον 600 εκατομμύρια για το GovSatcom και άλλα 600 για το SSA. Όσον αφορά το συνολικό πλαίσιο, Βεβαίως όλη η εργασία που κάνουμε οπωσδήποτε έχει σαν στόχο να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα ε, στα ιστορικά παραδοσιακά προγράμματα, τα οποία πρέπει να ενδυναμωθούν όσο γίνεται περισσότερο, ο Γαλιλαίος και ο Κοπέρνικος οπωσδήποτε. Αυτά ήθελα να σας πω και ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ε, ότι η πρώτη ε, δημοσίευση του προγράμματος έγινε τον Ιούλιο. Από τότε ε, οι διεργασίες για το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ εντατικές. Είπατε κι εσείς ότι υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες. Έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας. Πρέπει να περάσουμε Συνεπώς ευθύ αμέσω ε, κατόπιν της εισαγωγή ε, από τον εισηγητή στους σκιώδεις εισηγητές ή ε, σε όσους τους αντικαθιστούν. Δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Κυρία Μουντε. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι αντικαθιστώ την Κωνσταντζα Κρέλ, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ Ξέρω όμω ότι έχει συνεργαστεί πολύ καλά με τον εισηγητή και τον ευχαριστεί για τη δουλειά του. Η εστίαση της, ε, τροπολογία, των τροπολογιών της ε, Κωνσταντσα είναι, αφορούν καταρχάς την ασφάλεια και την άμυνα γιατί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δίνουν μια νέα βαρύτητη, βαρύτητα σε αυτό το θέμα. Επίση, η ομάδα μα πάντοτε θεωρούσε ότι το διαστημικό πρόγραμμα πρέπει να παραμείνει πολιτικό και οι συμπράξει με τον τομέα τη ασφάλεια είναι πραγματικότητα, αλλά θέλουμε να, υπάρχει αυτή, ε, να μην υπάρχει αυτός εστίαση ε, του προγράμματο του διαστημικού, όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ε, η πρόσληψη, το πώ το καταλαβαίνουν οι χρήστε, το έγνο και το γαλιλαίο, πρέπει να ενισχύσει ε, δεν έχουμε επαρκή αποτελέσματα ε, και όσα γνωρίζουμε δεν είναι ικανοποιητικά. Επομένως θέλουμε να δοθεί μεγαλύτερη ευθύνη στο GSA ε, που έχει άμεση σχέση με τον τελικό χρήστη Όσον αφορά τώρα τις προτάσεις COFSATCOM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα έχει προστιθέμενη αξία. Τα κράτη-μέλη διαφωνούν για την αναγκαιότητα επιπλέον ε, ε, ικανοτήτων και ο προπολογισμό είναι πολύ περιορισμένος για να επιτευχθούν όλα αυτά, οπότε η ε, συνάδελφος προτείνει να διαγραφούν οι προτάσεις ε, της GovSatcom για να μπορέσει να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός ε, σε, ε, στην ενίσχυση δορυφόρων ώστε να μην κινδυνεύουν τα έγνος και γαλιλαίο. Βεβαίως ε, είμαστε υπέρ του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου. Επίσης ε, υπάρχει ασυμφωνία όσον αφορά την εστίαση στους τελικούς χρήστες, δηλαδή ο GSA πρέπει να έχει περισσότερους, ε, περισσότερες ευθύνες. Το θέμα των δημοσίων προμηθειών και το άνοιγμα σε περισσότερους φορείς συζητείται τώρα. Επόμενο στάδιο να συζητήσουμε τους γενικότερους στόχους πριν μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και είμαστε πεπισμένοι σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα ισχυρό κείμενο για το διαστημικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι κατάλληλο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες της. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά στον κύριο Χένκελ, αντί του κυρίου Τοσανόφσκι που δεν είναι παρόν. Ευχαριστώ. Και να πω καταρχάς ότι προτείνει πιο ενισχυμένο ρόλο της υπηρεσία και μεγάλη δυνατότητα μεταφοράς με το Γαλιλαίο. Και άλλα προγράμματα θα πρέπει να υποφελούνται από τις συνεργίες και από την εμπροκνομοσύνη της Υπηρεσία. Και επίσης αυτόνομη ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει σεβαστή από τα κράτη-μέλη. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό και τους συντελεστέ, ως και μας πιστεύει ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα στο να υπάρχει η υπηρεσία αυτή, αλλά ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια υπηρεσία επικοινωνίας με τις κυβερνήσεις και σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και την υποπτία του διαστήματος θα πρέπει να αυξηθούν τα χαρτοφυλάκια και τα κοντήλια, όπως είπαν οι συνάδελφοι, όχι εις βάρος του Γαλιλαίου και του Κοπέρνικους. Και τέλος, η συμμετοχή των τρίτων χωρών. Είμαστε πεπισμένοι ότι η συμμετοχή κάποιων χωρών, όπως η Βρετανία μετά τον Brexit, είναι προς το συμφέρον καταρχάς της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα είμαστε αντίθετοι με τις πολιτικές και τους σκοπούς του κυρίου Μπαρνιέ που θέλει να τους αποκλείσει. Οι διεθνείς λοιπόν συμφωνίες θα πρέπει να επιτρέπουν στις τρίτες χώρες να συμμετέχουν στα προγράμματα συμπεριλαμβανομένων και του προγράμματος γαλλιλαίου και του προγράμματος Έγνωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λοιπόν Πρόεδρος. Τρίτος. Η κυρία Ναχτογάλα. Yes, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σαλίνη για τη δουλειά που έκανε. Και οι υπόλοιποι το πρόγραμμα για το διάστημα θεωρώ ότι συνενώνει τις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που ήδη υπάρχουν. Συμφωνώ με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το πρόγραμμα έχει δυνατότητα υποστήριξη της καινοτομίας αλλά και τις οικονομικές δραστηριότητες στους τομείς downstream. και την συνολική οικονομία και επίσης τις δυνατότητές μας παρακολούθησης του κλίματος, το οποίο αποτελεί ένα τμήμα της πρόταση το οποίο καλωσορίζω. Και αυτό περιλαμβάνει και ένα στοιχείο που έχουν σαφή και έχει σαφή προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει μεγάλες ευκαιρίες για την ε, εναρμόνιση των προγραμμάτων αυτών και τη δημιουργία νέων συνεργείων. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι υπέρ μαζί με τον σκιώδη και τον, σκι... με τον εισηγητή και τον σκιώδη υπέρ των προτάσεων αυτών που έχουν καταθέσει. Έχω και κάποιες ε, αμφιβολίες ωστόσο σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ε, Διαχειριστική Επιτροπή. Πολύ φοβάμαι ότι η διαδικασία διοργάνωση διαγωνισμών θα δυσκολέψει έτσι περαιτέρω. Δεν θα απλοποιηθεί. Και νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε όλε αυτέ οι αλλαγέ να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τη διαδικασία. Για τον ορίζοντα 2 τη Ευρώπη τώρα, Horizon Europe. Πιστεύω ότι το τμήμα για το διάστημα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και τονίζω τις συνέργειες μεταξύ προγράμματος διαστήματος και Horizon Europe. Τέλος, τελευταία ανησυχία που θα ήθελα να εκφράσω. Σε ό,τι αφορά την προσθήκη νέων συντελεστών στο πρόγραμμα, πιστεύω ακράδαντα ότι καταρχάς θα πρέπει να φροντίσουμε τη συνέχεια του προγράμματος και των υπόλοιπων flagship προτού ξεκινήσουμε να αναπτύσσουμε νέα τέτοια προγράμματα. Ιδιαίτερο δεδομένου ότι από τη φαίνεται δεν έχουμε τα χρήματα να συντηρήσουμε τους παλιούς συντελεστέ. Δεδομένων όλων αυτών λοιπόν πρέπει να πω ότι προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδες. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Η πράσινη. Είναι εδώ ο κύριος Γιάκουρο. Όχι. Άρα ήρθε η σειρά μου, γιατί και εγώ σκιώδης είμαι από την ΚΟΥΑ. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Τα προγράμματα λοιπόν για το διάστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι τρέχουσες, οι υφιστάμενες υποδομές ως προς τους δορυφόρους με πιο εμβρία χρήση των προγραμμάτων αυτών. Έχουμε ήδη αναπτύξει ένα, το Γαλιλαίο, άλλο ένα, τον Κοπέρνικο. Και φυσικά είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε όχι γενικά και αόριστα μόνο το ρυθμό των εξελίξεων στα περιβαλλοντικά θέματα κτλ. Αλλά και λεπτομερώς να εξετάσουμε τον αντίκτυπο της αύξησης θερμοκρασίας, της ξηρασίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε χώρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές επιπτώσεις για την αρχαιολογία, για παράδειγμα, στην περίοδο της ξηρασίας. Φυσικά, είμαστε κατά της διτής χρήσης τμήματων κάποιων προγραμμάτων και είμαστε ιδιαίτερως κατά του να αντιτεθούν όλα τα χρήματα στον Καλλιλέο GSA και τον Κοπέρνικο. Όπου εισαγάγονται νέοι συντελεστές στα προγράμματα, θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχα ε, νέα τμήματα του προϋπολογισμού, που θα τους εκπληρωθούν ιδάλλως θα διακυβευτούν τα πολύ καλά και θετικά αποτελέσματα σημαντικών τμήματων του προγράμματος. Θεωρώ λοιπόν ότι επαρκούν τα σχόλια αυτά. Δεν ξεπέρασα μάλλον και τα δύο λεπτά και να δώσω το λόγο στον κύριο Ταμπουράνο. Grazie Presidente. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti per... Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ τον συνάδελφο ε, εισηγητή για την εξαιρετική εργασία του. Ε, είναι πολλά τα θετικά στοιχεία τα οποία μπορούμε να υποστηρίξουμε και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχει ευέλικτες και καινοτόμες δομές η Ευρώπη με ε, την δυνατότητα αυτόνομης προσέγγισης και πρόσβασης στο διάστημα. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες οι οποίες ευελπιστώ ότι θα ε, υπογραμμίσουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να καλύπτει ή καλύπτει ελλιπώς το κείμενο. Ε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία ζητούμε να δουν με προσοχή και οι συνάδελφοι και ο, εισηγητές, ο εισηγητής. Ο Κοπέρνικος ε, είναι σημαντικό για να γνωρίζουμε ε, τι συμβαίνει στην επικράτειά μας. Το στοιχείο για μας αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε με περισσότερα, ε, περισσότερους πόρους αλλά και με περισσότερες δυνατότητες. Κυρίως όσον αφορά την μελέτη των μετεωρολογικών κερικών καιρικών φαινομένων, ε, της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής κλπ. Επίσης πιστεύουμε ότι ο Κοπέρνικος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα παρατήρησης της πολιτιστική κληρονομιά, όπως άλλωστε ανέφερε και η σκέδωση συγγήτρια τη ε, ΓΚΟΕ. Ε, αλλά πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να μελετά διαρκώ την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υποδομέ της χώρε μέλη ε, επίσης ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να δούμε τις πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες κινούνται στον τομέα αυτό και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να πιστοποιηθούν οι διαστημικές υπηρεσίες και αυτού του είδους οι διαδικασίες. Διαφάνεια. Είναι πολύ σημαντικό, ε, έστω και αν το αναφέρω τελευταίο, ε, να αναφερθούμε στην διαφάνεια. Μεγαλύτερη διαφάνεια. Ε, θα πρέπει, ας πούμε, να, υπάρχει, να δημιουργηθεί ένα είδος φόρουμ χρηστών. Θα πρέπει οπωσδήποτε μέσω αυτών των στοιχείων να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές λειτουργικές, τωρινές και μελλοντικές ανάγκες του συστήματος και επομένως να λειτουργήσει σωστά το σύστημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Συνάδελφε συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της DigiGrow. Grow. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή κύριο Σαλίνη για την έκθεσή του, η οποία κατά την άποψή μα ταυτοποιεί τα πιο σημαντικά στοιχεία της προτάσεως τη Κομισιόν. Δηλαδή υπογραμμίζει την σημασία ε, της διαστημικής ε, οικονομίας που αποτελεί μεγάλη οικονομική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης καθορίζει σωστά και περιγράφει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την διακυβέρνηση. Επίσης, ε, όπως και ο εισηγητής και εμείς θεωρούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να αποφευθούν οι επικαλύψεις. Επαναλαμβάνουμε ότι η ανάγκη ε, αποσαφήνισης με ένα και μόνο Financial Partnership Framework ε, ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ε, σωστή υλοποίηση του προγράμματος μέσω της υπηρεσίας στο Παρίσι και της άλλης στην Πράγα έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τον ρόλο των διαφόρων φορέων που θα είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των προγραμμάτων και ε, η υπηρεσία του Παρισιού και ο οργανισμός της Πάγας ε, θα πρέπει να είναι η μόνη υπεύθυνη για την υλοποίηση ε, του προγράμματος και την χρήση του προϋπολογισμού. Όσον αφορά δε τον προϋπολογισμό, σωστά ο εισηγητής αναφέρεται στον προϋπολογισμό. Για πρώτη φορά όμως υπενθυμίζω ότι η Κομισιόν αποδίδει μεγάλη σημασία στον Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο αλλά ταυτόχρονα προτείνει και ενδεικτικά ποσά τα οποία σιγά σιγά ε, θα επιτρέψουν καλύτερη διαχείριση και θα δοθεί η δυνατότητα ε, να χρησιμοποιηθούν σωστά τα κονδύλια ακόμα και να αυξηθούν ε, τα κονδύλια. Κατανοούμε την πρόταση της έκθεσης για αύξηση του προβλεπόμενου ποσού θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονό ότι πρόκειται για δύο προγράμματα τα οποία βασίζονται σε υφιστάμενες υποδομές σε επίπεδο κρατών μελών και που ευνοούν ε, ε, επενδύσεις από την πλευρά των κρατών μελών. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ευελιξία όπως το ανέφερα ήδη, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα άμεσης συμμετοχής των κρατών μελών, διότι οι υποδομές που ήδη χρησιμοποιούνται σήμερα είναι οι υποδομές των κρατών μελών και επομένως ο εξυγχρονισμός τούτων των υποδομών ε, η επένδυση σε νέες υποδομές μπορεί να γίνει μέσα από συγχρηματοδοτήσεις εθνικές από την πλευρά των χωρών που ήδη έχουν και διαθέτουν τέτοιες υποδομές. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Όντως είναι σημαντικές οι προκλήσεις και τα διακυβεύματα. Βεβαίως εμείς την Ομενεβή σε όλες τις προτάσεις ε, τις οποίες το Κοινοβούλιο θα μπορούσε μέσω των διαφόρων πολιτικών ομάδων να υποβάλει. Πάντως να ξαναπούμε ότι πρόκειται για αστικό πρόγραμμα, ε, δηλαδή μη στρατιωτικό, ε, ε, ένα πρόγραμμα που αφορά μη στρατιωτικές υποδομές. Και βεβαίως οι ίδιες οι χώρες θα έχουν πλέον την ευθύνη της χρήσης σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για λόγους άμυνας. Αυτά, ε, ε, ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, η άποψη της Κομισιόν έτσι όπως την παρουσιάζει και στο Συμβούλιο και η θέση του Συμβουλίου έτσι όπως διαφαίνεται είναι πολύ κοντινή με την θέση που παρουσίασε σήμερα ο εισηγητής. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι σε διοργανικό επίπεδο θα καταφέρουμε ε, να επιτύχουμε σε ε, σωστό χρονοεύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την αρχή της επόμενης χρονιάς, καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εξαιρετικό αυτό που μας λέτε, ότι η Κομισιόν δηλαδή έχει την ίδια άποψη με μας. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Μετά και με τα μέλη της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να ξαναδώσω τον ε, ε, λόγο ε, για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση στον εισηγητή, τον κύριο Σαλίνη. Κύριε Σαλίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια θα πω μόνο. Ξεκινώ από την τελευταία σκέψη ε, της Κομισιόν που υπογράμμισε κάποια στοιχεία τα οποία, στα οποία αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι στις παρεμβάσεις τους. Ε, μία από τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος, είναι ότι πρόκειται ένα μη στρατιωτικό πρόγραμμα και θέλουμε να παραμείνει μη στρατιωτικό αλλά θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν ακριβώς τη φύση του όσο γίνεται περισσότερο. Μιλάμε επομένως ε, για υπηρεσίες, ε, για βιομηχανία, ε, το θέμα της κυβερνοασφάλειας κλπ. Στοιχεία λοιπόν τα οποία αφορούν καθαρά μη στρατιωτικό πλαίσιο. Ε, και βεβαίως μπορεί να έχει και ένα παρακλάδι ε, που θα αφορά την άμυνα, αλλά ο πυλώνας επί του οποίου βασίζεται δεν είναι η άμυνα, είναι ακριβώς ε, όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως, τα μη στρατιωτικά. Εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η σχέση με την βιομηχανία και αυτό μας είναι ιδιαίτερος προσφυλής ως ιδέα. Να πω κάτι που ξέχασα στην εισαγωγή μου. Το θέμα του Horizon Europe, Horizon Ευρώπη, είναι απαραίτητο να ε, ε, βάλουμε όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν από το διαστημικό πρόγραμμα στον ορίζοντα Ευρώπη, ε, στο κεφάλαιο που θα αφορά την έρευνα, τη χρηματοδότηση της έρευνας για το διάστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο, το θέμα του προϋπολογισμού και της ευελιξίας του προϋπολογισμού στο εσωτερικό του. Ε, ζητούμε λοιπόν από την Κομισιόν να μην ε, έχει άκαμπτα όρια όσον αφορά τον προϋπολογισμό που έχει δοθεί ε, στα διάφορα στοιχεία και το γεγονός ότι το ανέφερε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Τέλος, να ξαναευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους. Θεωρώ ότι υπάρχουν όλες ε, οι ε, απαραίτητες προϋποθέσεις για μια διαπραγμάτευση σωστή και όχι πολύ μακροσκελή. Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα έχετε την δυνατότητα και την ευκαιρία να συζητήσετε όμορφα και καλά όλες τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το επόμενο. So, as agreed... Όπως συμφωνήσαμε, το δεύτερο σημείο στο στην ημερήσια διατάξη μα θα είναι η πρόταση του κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματο συνδρομή στον παροπλισμό του Περινόηλεκτρικού ηλεκτρικού σταθμού Ιγναλίνα στη Λιθουανία. Πρόγραμμα Ιγναλίνα και για την κατάρτιση του κανονισμού 1369 του 2013. Είναι. I would Να σας υπενθυμίσω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει να κάνει με το πρόγραμμα παροχής υποστήριξης για τον παραπλήσμα του πυρηνού ηλεκτρονικού σταθμού Ιγνάλινα στη Λιθουανία και για τον προπολογισμό περίοδο 2021 έως 2017. Δεν χρειάζεται διαβούλευση με το Κοινοβούλιο επισήμω, αλλά το Συμβούλιο αποφάσισε να διαβουλευτεί με το Κοινοβούλιο. Άρα, συνάδελφοι, συζητάμε το θέμα δύο αντιδραστήρων και όλες τι σχετικέ υποδομέ. Η, η Επιτροπή Ήτρε είναι η καθήλυνα αρμόδια και η Επιτροπή Budget δεν θα γνωμοδοτήσει. Έτσι αποφάσισε. Άρα, στα χέρια μα είναι το θέμα αυτό. Και κύριο ε, Γιάνβουρ θα πάρει το λόγο εξ ονόματο τη κυρία Χάρμ και θα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση το οποίο συναποτελείται από 18 18 τροπολογίες. Έχουμε 20 λεπτά για τη συζήτηση. Γι' αυτό σας παρακαλώ να επικεντρωθείτε στα πιο βασικά. Οι σκιώδεις θα έχουν 2 λεπτά στη διάθεσή τους και οι υπόλοιποι από ένα λεπτό όπως προβλέπετε στις συνεδριάσεις ομάδος. Ο κύριος Γιάβορ λοιπόν έχει το λόγο και θα ξεκινήσει τη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αναφέρθηκε ότι θα έπαιρνε το λόγο εξ ονόματος της Ρεμπέκα Χράμς, η οποία ζητά συγγνώμη γιατί δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στη συζήτηση αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω της επίσκεψης που έχει αναλάβει στις ΕΠΑ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, εξω, ε, πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτιμάζοντας την έκθεση αυτή, εξέτασα ε, εντελεχώ την κατάσταση και συναντήθηκα με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς και τους ε, εργαζόμενους της Σιγναλίνα και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, της εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕΠ. Από τότε λοιπόν που παρακολουθώ εξ αρχής μάλλον το πρόγραμμα Εκναλίνα Έχω να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις εργασίες της και έχουν διορθωθεί τα παλαιότερα προβλήματα. Τα προβλήματα λοιπόν αυτά έχουν διαπιστωθεί από ανεξάρτητους εμπρογνώμονες και παρουσιάστηκε και από σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην έκθεσή μου αναφέρω δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε. Καταρχάς το θέμα τι σύγκνα είναι. Είναι πολύ ευρύ πρόγραμμα Έχουμε υπολογίσει λοιπόν το κόστος της, ε, του παροπλισμού και συμφωνούν και η ΕΤΕΠ και η κυβέρνηση της Λιθουανίας και οι προγνώμη της Λιθουανίας. Παρά όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει 552 εκατομμύρια για τον παραπλησμό καταρχάς της δεύτερης μονάδας που θα ξεκινήσει το 2026 και θα φτάσει μέχρι το 2027. Υπάρχει λοιπόν ε, μια χρηματοδότηση η οποία θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί πριν να ξεκινήσουν καν τα έργα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε 780 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό το τελευταίο αυτό ποσό να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει πίσω σε όχι αφορά τη δεσμεύσεις της για το πρόγραμμα Αγναλίνα εις βάρος της Λιθουανίας. Και η Λιθουανία και η συνεισφορά τη θα πρέπει να είναι κατά αναλογία των όσων προβλέπονται στα σχετικά πρωτόκολλα και στι συνθήκε προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω αυτό το πρόγραμμα, την έκθεση μάλλον, να την υποστηρίξουν και οι σκιώδει συζητητέ και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο, για τα εισαγωγικά αυτά σχόλια και νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικά της κατάστασης. Ο κύριος Λάγκεν καταρχάς από το ΕΛ. Πείτε. Σας ευχαριστώ. Είχε αλλάξει η ημερήσια διάταξη γιατί το θέμα αυτό το προβλέπαμε για αύριο νομίζω. Έχουμε ασχοληθεί επισταμένως και σε πολλές περιστάσεις με το πρόγραμμα Ιγναλίνα. Καταρχάς το 2006 το 2009 επίσης βάσει της ε, συνθήκης προσχώρησης πρόκειται για πυρηνικούς αντιδραστήρες ρωσικής κατασκευής. Ε, το επισκέφτηκα και εγώ τα, τις εγκαταστάσεις. Μιλάμε για τεράστιες εγκαταστάσεις, τεράστιες υποδομές. Το κόστος δε της ανοικοδόμησης είναι συνολικά 2,9 δισεκατομμύρια εκεί, σε αυτό το ύψος εκτιμάται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τα 2,4 δισεκατομμύρια και τώρα λοιπόν το θέμα είναι να υπάρξει μια λογική και ομαλή μετάβαση μεταξύ του παραπλησμού του πρώτου αντιδραστήρα και της θέση σε λειτουργία του δεύτερου αντιδραστήρα. Έτσι λοιπόν υπάρχει κάποιο νόημα όταν θα γίνει διακοπή βάσει του προηγούμενου δημοσιονομικού πλαισίου και από πλευρά προμηθειών και από πλευρά εξειδικευμένου προσωπικού, ενδεχομένω να υπάρχουν ε, επιπλέον ε, δαπάνε, επιπλέον κονδύλια που θα πρέπει να καλυφθούν πέρα από τα προβλεπόμενα. Γι' αυτό λοιπόν η προσέγγιση τη κυρία Χάρεμ σε ό,τι αφορά την κάλυψη του οικονομικού και δημοσιονομικού αυτού κενού πριν καν προκύψει είναι σωστή και κατάλληλη. Αλλά στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου είναι σαφές το τι ακριβώς μπορούμε να προβλέψουμε. Εμείς κάνουμε μία γνωμοδότηση, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ελέγχει και το 2012 ήδη είχε σχολιάσει με επικριτικό τρόπο η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του κατά πόσον ήταν σκόπιμες οι δαπάνε αυτέ. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες ελλαγές, κάποιε τροποποιήσει και τελικά καταφέραμε τουλάχιστον να ελέγξουμε λίγο το κόστος του πρώτου τουλάχιστον αντιδραστήρα. Για μένα, πέρα από τον παραπολισμό των αντιδραστήρων, το θέμα που τύφεται είναι το εξής. Η... Τα καύσιμα έχουν ήδη αφαιρεθεί. Είναι σε μια ανοιχτή αποθήκη 10 χιλιόμετρα από την Ιγναλίνα και ως εκ τούτου θα χρειαστεί, σύμφωνα με όλους τους υπολογισμούς, αυτό το σχετικά α, μη ασφαλή χώρα αποθήκευση να το συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσον στα πλαίσια των προγραμμάτων υπάρχει δυνατότητα αυτή η ανοιχτή αποθετευτική χώρη να ληφθούν υπόψη και να συμπεριληφθούν στους χώρους ε, που είναι υπό και εγώ έχω επισκεφτεί 4-5 φορές ε, τις εγκαταστάσεις οι ε, Ρώσοι λοιπόν επιχειρηματία ε, την πρώτη φορά, συγγνώμη, ε, μα, οι Ρώσοι εμπειρογνώμονε είχαν πει ότι μετά την πρώτη δαπάνη των 300 εκατομμυρίων δεν υπήρχαν περιθώρια, δεν υπήρχαν κίνδυνοι ατυχήματο. Και μετά το Τσέρνομπιλ λοιπόν έχει καθοριστεί και μια διαδικασία κατά την οποία όχι μόνο γίνονται έλεγχοι εκ των υστέρων, και σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις ε, των τιμών ενέργειας που θα προκληθούν ε, από τον παραπλήσμο του αντιδραστήρα αυτή. Είναι δύσκολο λοιπόν το πρόγραμμα. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της συνεχιζόμενης ε, χρηματοδότησης. Δίκιο έχετε, λέει ο Πρόεδρος. Όταν κάποιον τον έχουμε αναγκάσει να κάνει κάτι, θα πρέπει τουλάχιστον να καλύψουμε το κόστος του δημοσιονομικό. Επόμενος, ο κύριος Γκρούμπασεφ. Σκιώδης από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υποστηρίζω την έκθεση της Ρεμπέκα Χάμς, ε, ειδικότερα όσον αφορά την ενίσχυση του προγράμματος παροπλισμού. παροπλισμού. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε δεχόμαστε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι 350 εκατομμύρια, ή αν δεχτούμε την πρόταση της Λιθουανικής Κυβέρνησης που είναι 750 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν άκουσα την άποψη της Επιτροπής Προπολογισμών για αλλαγή αυτού του ποσού. Από την άλλη υπάρχει μία πρόταση για την αύξηση του, ε, ποσού για την Βουλγαρία ε, και την Τσεχία που δεν ε, χρειαζόταν. Οπότε δεν καταλαβαίνω. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς την κυρία Χάρμ. Στο πρώτο ερώτημα για το εξειδικευμένο προσωπικό, τι ακριβώς προσωπικό. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει αυτή Ε, είπατε ότι χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ενημέρωση στο πλαίσιο του προγράμματος ε, παροπλισμού διαφορετικά πρέπει να καλύπτεται από τον κανονισμό. Θα έπρεπε να υπάρχει και μία αξιολόγηση του πώς η χρηματοδότηση της Ένωσης για τον παροπλισμό θα έχει αντίκτυπο στην περιοχή, ειδικότερα όσον αφορά ε, στο προσωπικό ε, και τους ειδικού που εργάζονται για τον παροπλισμό. Για την 14 τροπολογία, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλετε θέλει να επιτύχει και τη διάδοση του, ε, της πληροφορίας που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει αρκετή γνώση όσον αφορά τον παροπλισμό τέτοιου είδους αντιδραστήριων. Ίσως θα έπρεπε να γίνει μια καλύτερη χρήση ε, των κονδυλίων που υπάρχουν για τις δραστηριότητες του παροπλισμού. Κάτι ακόμη δεν είναι ακριβώς ρωσικού τύπου αντιδραστήρες, γιατί υπάρχουν πολλά είδη είναι αυτό ακριβώς το RBM, το RBMK που χρησιμοποιεί το Σοβιετική Ένωση στη Σλοβακία και την Τσεχία είναι διαφορετικού είδους, είναι 440 και σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτές τις χώρες και τον παροπλισμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη Λιθουανία, γι' αυτό χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται περαιτέρω χρηματοδότηση 780 και όχι 750 εκατομμυρίων ευρώ για να αρχίσουν να εργάζονται σε αυτήν την επτάετη περίοδο, όχι μόνο μόνο να την τελειώσουν, το κομμάτι που αφορά το πρώτο αντιδραστήρα, αλλά να συνεχίσουν και το δεύτερο αντιδραστήρα. Αν το αναβάλουμε, μετά θα αρχίσουμε να συζητούμε τι θα κάνουμε για το δεύτερο αντιδραστήρα και δεν νομίζω ότι ε, τα έργα για το δεύτερο αντιδραστήρα πρέπει να περιμένουν την ολοκλήρωση των έργων του πρώτου αντιδραστήρα. Νομίζω ότι αυτέ οι δύο εργασίε πρέπει να γίνουν παράλληλα. Διαφορετικά, ο χρονικό μα ορίζοντα θα φτάσει το 2040 ενδεχομένω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το θέμα του καυσίμου. Εντάξει, το καύσιμο μπορούμε να το απομακρύνουμε. Το πρόβλημα είναι ο γραφίτης που χρησιμοποιείται στην αντίδραση, γιατί υπάρχει πολλής γραφίτης σε μεγάλη συγκέντρωση και είναι πάρα πολύ δύσκολο και το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα αφαιρεθεί αυτός ο γραφίτης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει υπό τον GRC μία ομάδα παροπλισμού που θα μπορέσει να συλλέξει εμπειρίες από τις διάφορες χώρες και από διάφορα ίδρια αντιδραστήρων για να χρησιμοποιηθεί αυτή η γνώση για το μέλλον, για τον μελλοντικό παροπλισμό διαφόρων ειδών αντιδραστήρων. Απλώς για να γνωρίζετε Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι 39 αντιδραστήρες με γραφίτι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας το λέω απλώ για να το γνωρίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Σε γενικές γραμμές υποστηρίζω την έκθεση ε, της ε, Ρεμπέκα Χάρμς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές οι παρατηρήσεις που κάνατε. ECR δεν εκπροσωπείται σε επίπεδο σκιωδών. Ε, τώρα η φιλελεύθερη λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, ως άλλη θα θέλαμε πρώτα να ευχαριστήσουμε την ε, Ρεμπέκα για τη βαθιά γνώση του θέματος που έχει. Μίλησα μαζί της και επιβεβαιώνουμε ότι είναι κοινή λογική τα όσα λέει. Και η αιτιολόγηση που δίνει στην έκθεσή της με βρίσκει σύμφωνους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί ε, εάν δεν υποστηριχτεί η χρηματοδότηση δεν θα γίνει, δυνατή, ε, δεν θα γίνει δυνατός ο παροπλισμός στην ε, κατάλληλη προβλεπόμενη περίοδο. Επίσης θα δημιουργούσε πρόβλημα ε, στις, ε, ε, στην τεχνογνωσία που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι και οι ομάδες οι οποίες ασχολούνται με το ζήτημα αυτό. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική η θέση που κάνει η συγγήτρια ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια θα πρέπει να αφορούν τον παροπλισμό του αντιδραστήρα και όχι ε, άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε ε, σπατάληση του χρήματος. Τούτων λεχθέντων έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες ως άλντε και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις άλλων ε, μελών, αλλά ε, ακολουθούν οι τροποποιήσεις τροπολογίες μας κάποιες ε, κάποιες αρχές. Πρώτον, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν παραπάνω, α, ότι υπάρχουν ε, περίπου 90 ε, που πρέπει να παραπληστούν και μόνο στη Γερμανία έχουν παραπληστεί 5 οι δαπάνες του παροπλισμού οπωσδήποτε θα αποτελέσουν εχμή του δόρατος στους προϋπολογισμούς πολλών χωρών. Επίσης, η Άλντε θεωρεί ότι δεν θα πρέπει ε, η περίπτωση της Λιθουανίας, της Βουλγαρίας ή της Σλοβακίας να θεωρηθούν ως ε, προηγούμενα, έτσι ώστε να θεωρηθεί υποχρεωτική η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε μελλοντικές ε, παροπλιστικές διαδικασίες. Τέλος. Θα υποβάλουμε τροπολογίες έτσι ώστε να συζητηθούν άλλες ε, πιθανότητες, δυνατότητες χρηματοδότησης εναλλακτικά προς τον ευρωπαϊκό ε, ε, προϋπολογισμό όσον αφορά την, τον παροπλισμό των αντιδραστήρων. Δηλαδή να μην υπάρχει μόνο αυτή και μόνο η δυνατότητα. αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πίεζε πάρα πολύ κάποιο κράτος μέλος να κλείσει έναν αντιδραστήρα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η χώρα μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τον παροπλισμό. Αν η Γερμανία, για παράδειγμα, αποφάσισε να παροπλήσει σταδιακά δεκάδες αντιδραστήρες. Αυτό είναι μεγάλο κόστος. Ε, βέβαια αυτό είναι και μια ανεξάρτητη εθνική, εθνική τους απόφαση. Το ίδιο ισχύει και με τη Γαλλία, με, κάποιους, ε, με κάποιες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Είναι καθήκον τους. Αν όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαναγκάσει, εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής, οπότε έχω και εγώ δύο λεπτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εξανάγκασε οποιοδήποτε κράτος υποψήφιο για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παροπλήσει ένα ένα αντιδραστήρα, τότε πρέπει να υπάρχει και η απαραίτητη χρηματοδότηση. Ένα ζήτημα είναι τι θα κάνουμε με το γραφίτι, γιατί αυτό είναι ένα είδο αντιδραστήρα που, χρησιμοποιούν το γραφίτι, που χρησιμοποιεί το γραφίτι. Και κάτι ακόμη είναι τι θα γίνει με το καύσιμο γιατί υπάρχει πάντοτε ουράνιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να τύχει νέα επεξεργασίας ε, κλπ. Τρίτο σημείο, Επίσης υπάρχει χαμηλής ραδιενέργειας ε, ε, τσιμέντο. Οπότε το θέμα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η τεράστια διαφορά μεταξύ 700 και 400, συγγνώμη, 450 και 780 εκατομμυρίων ευρώ ε, θα καλυφθεί. Ολοκληρώνουμε λοιπόν για το σημείο αυτό λέγοντας ότι πρέπει να αποφασίσουμε μέχρι κάποια χρονική στιγμή μπορούμε να υποβάλουμε τις τροπολογίες μας και μετά πολύ σκληρή θα είναι η δουλειά της ε, Ρεμπέκα Χάρμς να δει πώς θα συγκεράσει όλες αυτές τις τροπολογίες σε μία σαφή πρόταση. Λοιπόν, μετά τους σκιώδεις εισηγητέ, να δώσω τώρα το λόγο σε άλλους συναδέλφους και ερώπε. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να πω το εξή. Τα έγγραφα αυτά, όπως η γνωμοδότηση της Ρεμπέκα, κάνουν τους Ευρωπαίους πολίτες να πιστεύουν σε μας, να πιστεύουν στο ευρωπαϊκό αυτό έργο. Χαίρομαι λοιπόν που υποστηρίζετε και από την Επιτροπή μας και από το Κοινοβούλιο. Από την άλλη, αν απορρευθούν οι τροπολογίες, το σοκ θα είναι τεράστιο για τους πολίτες της Λιθουανίας. Πολύ απλά θα πιστέψουν ότι η Ευρώπη υπαναχωρεί σε σχέση με τις ε, δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και τις υποσχέσεις της. και ότι δεν επιθυμεί πλέον, δεν έχει πρόθεση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ε, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να σα επιστήσω την προσοχή και σε κάτι άλλο, σε ένα άλλο ε, εντονότατο πρόβλημα που έχει να κάνει με τον ε, παροπλισμό του σταθμού Ιγναλίνα. Δεν δίδεται από το 2008 και μετά υποστήριξη προς τη γενικότερη περιοχή, γιατί ο παραπλησμός προφανώς έχει επηρεάσει πάρα πολύ και τη συνολική περιοχή. Υπάρχει μια ολόκληρη κομμόπολη, 35.000 άτομα, οι οποία συντηρούνταν από τον ε, πυρηνο ηλεκτρικό σταθμό και πλέον μαστίζεται από τα πιο υψηλά <coughs> ποσοστά ανεργίας. Επίσης, είναι αποτελείται από πολλές μειονότητες που είχαν συγκεντρωθεί για τη συντήρηση του σταθμού. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν για την ανάπτυξη της ε, περιοχής αυτής και να εκπληρώσουμε τη συνθήκη παριθμών, την συνθήκη και το πρωτόκολλο 4. Ελπίζουμε λοιπόν οι κοινωνικοί δείκτες της περιοχής αυτής να φτάσουν στο μέσο όρο τουλάχιστον της Λιθουανίας. Όπως είπε και ο κύριος Λάνια από τη Γερμανία, το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζουμε την προσωρινή μόνο αποθήκευση των καυσίμων. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και αυτό δεν έχει ξεκινήσει καν ως θέμα. Μιλάμε για μια πεντακονταετία αποθήκευσης. Η Λιθουανία λοιπόν χρησιμεύει, χρησιμοποιούσε μάλλον τον σταθμό αυτό για το 20% της παραγωγής ενέργειας της. Ήταν ε, σοβιετική, σοβιετικό κλειδοδότημα και τώρα φυσικά η Λιθουανία έχει μείνει με όλες τις συνέπειες του σταθμού αυτού, παρά το γεγονός ότι δεν αξιοποιούταν ιδιαίτερα. Αν το έργο αυτό εγκαταλειφθεί, θα φύγουν και όλοι οι μπρεγνώμονε και θα γίνει ακόμα πιο ακριβό το έργο αυτό. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε όσο πιο γρήγοροι και αποτελεσματικοί γίνεται. Και να φροντίσουμε να είναι όσο λιγότερο ακριβό γίνεται το έργο αυτό. Ε, εξετάσαμε και το ενδεχόμενο εξωτερική ανάθεση και τελικά προέκυψε ότι οι εταιρείε αυτέ που θα αναλάμβαναν ενδεχομένο στον παραπλησμό δεν ήταν σε θέση να διευθύνουν όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ο πρώτος αντιδραστήρας τέτοιου τύπου σε όλο τον κόσμο που θα χρειαστεί να παροπλιστεί και δεν ε, έχουμε υπόψη μας τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Θα είναι τεράστιος ο όγκος της εργασίας και θα πρέπει ενδεχομένω να μας βοηθήσουν και άλλες χώρες. Υποστηρίζοντας λοιπόν το σχέδιο έκθεση της ε, κυρία Χάρμς, ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε και τους όρους για περαιτέρω προγράμματα παροπλισμούς χωρίς επιπλέον κόστος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, από πλευρά σα. και θα θέλαμε τώρα να δώσω το λόγο στο Μάσιμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, αγαπητοί βουλευτές και θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους κοιότε για την προετοιμασία της έκθεσης. Είχα την χαρά να μεταβώ τον Ιούλιο μαζί με την κυρία Χάρμ στην Ιγναλίνα και νομίζω ότι η δουλειά μα ήταν ε, λεπτομερέστατη. Να σας υπενθυμίσω κάποια πράγματα και μετά να σας εξηγήσω γιατί καταβλήθηκε ή υποβλήθηκε μάλλον η πρόταση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 550 εκατομμύρια. Καταρχάς, η αρρωγή στο όλο πρόγραμμα παροπλισμού μέχρι τα τέλη του 2020, λαμβάνοντα υπόψη αυτή την επιπλέον πρόσταση ε, χρηματοδότηση, θα φτάσει τα 1,9 δι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο γεγονό είναι ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό μεταξύ των χρημάτων που χρειάζονται για να χρηματοδοτηθεί όλη τη δικασία μέχρι το 2038 και να γνωρίζετε και από την Λιθουανία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα φτάσει αυτό τα 1,33 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, το τρίτο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Πράγματι, ο παροπλισμός τέτοιου είδους αντιδραστήρων και τονίστηκε από πολλούς βουλευτές στη συζήτηση αυτή είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Πρώτη φορά συμβαίνει. Πρόκειται λοιπόν για μια επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να υιοθετήσει μια πολύ βαθμιαία και πολύ προσεκτική προσέγγιση. Το πρώτο λοιπόν βήμα θα είναι να γίνει μια μελέτη των υφιστάμενων ε, λύσεων για να δούμε πώ ακριβώ θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτόγνωρη επιχείρηση. Τα αποτελέσματα λοιπόν θα δημοσιευθούν μέχρι τα τέλη του 2021 μέσα 2022. Να σας το θέσω λοιπόν ως εξής υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες για το κατά πόσο γνωρίζουμε τι να κάνουμε καν στα πλαίσια του παροπλισμού. Γι' αυτό λοιπόν η βάση της χρηματοδότησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι το πρόγραμμα παροπλισμού, το οποίο συμφωνηθήκε το 2014 από κοινού με τον σταθμό Ιγναλίνα και με τις αρχές της Λιθουανίας, και γι' αυτό η συγχύτρια και ο εκπρόσωπος της, ο κύριος Γιάβορ, δήλωσε ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία για τη βάση του υπολογισμού αυτού. Αυτή η διαφορά λοιπόν οφείλεται στο κατά πόσο θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τον παροπλισμό του δεύτερου αντιδραστήρα μέσα στο πού αυτό ή στο επόμενο που Το τρέχον σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι ο δεύτερος αντιδραστήρας δεν θα παροπληστεί εκ παραλλήλου, αλλά μετά τον δεύτερο, την δεύτερη μονάδα και θα ξεκινήσει μετά το 2028. Στο επόμενο, πού το Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει τη χρηματοδότηση που θα επαρκεί και θα καλύπτει τις ανάγκες των τρέχων που Που Και παρεπιπτόντος είναι ήδη 20% πάνω από το ποσοστό που προβλεπόταν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Να σας υπενθυμίσω επίσης γιατί το ανέφερε και η συγκεντρία... ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν το ποσοστό χρηματοδότησης από 40% από τα 14% συγγνώμη, σε 20% στην ερχόμενη προγραμματική περίοδο. Να σας υπενθυμίσω εν είδη συγκρίσεως ότι σε σχέση με τα άλλα που λαμβάνουν σχετική οικονομική ενίσχυση βάσει των συμφωνιών που έγιναν στη Συμφωνία Προσχώρησης, Σλοβακία, Βουλγαρία, θα τα συζητήσουμε αυτά αύριο, συνεισφέρουν με ποσοστό 30 έως 40% με πολύ πιο υψηλό ποσοστό από αυτό που προβλέπετε για την ε, Λιθουανία. Αυτό μετά την έκθεση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, την ειδική έκθεση μετά από την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου το 2016. Ευχαριστώ πολύ. Thank you Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε λοιπόν τώρα γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη συνοχής γιατί ακριβώς ε, οι, οι οικονομολόγοι δεν μπορούν να αξιολογήσουν την κατάσταση επιτόπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ και τους κοιόδης εισηγητές ε, για όλες αυτές τις παρατηρήσεις επί της εκθέσεώς μου. Υπήρχαν κάποια πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία μπορούν να απαντηθούν ε, από την εισηγήτρια, τη Ρεμπέκα Χάρμς, αλλά θα ήθελα και εγώ ήδη να κάνω κάποια πρώτα σχόλια. Καταρχάς, όπως ε, υπόθηκε από πολλούς και ηγητές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόβλημα ε, στην καρδιά του προγράμματος είναι ότι ο χρονικός ορίζοντας ε, του προγράμματος παροπλισμός υπερβαίνει το επόμενο πι. Και γι' αυτό Εντάξει, κανένας δεν αμφισβητεί το συνολικό ποσό του, του παροπλισμού, 780 εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται για τον παροπλισμό. Το ζήτημα είναι πώς να πώς θα εξευρεθούν τα χρήματα γιατί πρέπει να υπάρξει μια χρηματοδότηση από το τρέχον πι και μετά ενδεχομένως και από το επόδημο. Δεν υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό το πι η οικονομική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί αυτό να έχει ως αποτέλεσμα ένα κενό ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο τμήμα της διαδικασίας της παροπλιστικής κάτι το οποίο μπορεί να αυξήσει και το κόστος παροπλισμού από οικονομικής καθαρά απόψεω έχει νόημα να διατεθούν τα χρήματα για ολόκληρη τη διαδικασία παροπλισμού ακόμη και αν η στην πράξη η δουλειά μπορεί να γίνει ακόμη και μετά το τέλος του επόμενου ΠΔΕΛΤΑΠΗ για να υπάρξει μια συνέχεια στο πρόγραμμα. Δεύτερο, ερώτημα, ε, δεύτερο ζήτημα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 14% της ίδιας συνεισφοράς ε, από τη Λιθουανία που θα αυξηθεί σε 20%. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια υπόθεση που είχε συμπεριληφθεί στην ε, συνθήκη προσχώρηση τη Λιθουανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα παροπλισμού τη Ιγναλίνα διέπεται από το πρωτόκολλο 4 της ε, Συνθήκης για την Προσχώρηση που δίνει τη δυνατότητα 100% ενωσιακής χρηματοδότησης για κάποια μέτρα και αυτό ήταν συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιθουανίας ότι 14% θα αναλάβει ε, ως προς το κόστος η ίδια η χώρα, κάτι το οποίο έχει γίνει ως τώρα και δεν βλέπουμε το λόγο να αλλάξει κάτι τέτοιο όπως είπε και ο συνάδελφος Ντένις Ρόπι ε, τέτοιου είδους αλλαγές ε, στις οριζόντιες δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να προκαλώσουν ενδεχομένω ε, κάποια ε, κακά αισθήματα στη χώρα που δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα τις παρατηρήσεις, η κυρία Πουνσέτη είπε για παράδειγμα ότι υπάρχουν και άλλες παροπλιστικές διαδικασίες ε, και δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όλες αυτές. Εντάξει, αλλά η Λιθουανία είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί στο επιχειρησιακό κόστος ε, που θα ε, δοθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είναι ένα τμήμα της, του ενεργειακού κόστους ε, και ε, είναι μια αξίωση του, των Ευρωπαίων φορολογωμένων πράγματι, αλλά νομίζω ότι η Λιθουανία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι δύο ξεχωριστά ζητήματα. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι συμφωνώ για τις υπόλοιπε πυρηνικές εγκαταστάσεις, η Λιθουανία όμως το είχε συμπεριλάβει στη συνθήκη προσχώρησής της και πιστεύουμε ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή η Λιθουανία κάνει πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες ε, οικονομικής φύσεως για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Και κάτι ακόμη, εξίσου σημαντικό, πολλοί σκιώδεις εισηγητές αναφέρθηκαν στη διάδοση της εμπειρίας από το πρόγραμμα Συμφωνώ Απολύτως. Ο παροπλισμός ε, θα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ε, στο ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά κατά τις επόμενες δεκαετίες. Υπάρχουν ήδη ε, δημόσιες συζητήσεις για την, τον παροπλισμό. γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πολύ καλύτερη επικοινωνία για τις παροπλιστικές διαδικασίες στην Ανατολική Ευρώπη. Όλες αυτές οι εμπειρίες πρέπει να γνωστοποιούνται ε, και ε, στις υπόλοιπες χώρες ε, που μπορεί να μην συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες αλλά ούτως ή άλλως σε επόμενες δεκαετίες πάρα πολλά κράτη-μέλη που έχουν πυρηνική ενέργεια θα βρεθούν σε μια αντίστοιχη κατάσταση και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει ένας ο καλύτερος δυνατός τρόπος παροπλισμού γι' αυτό ακριβώς συμφωνώ απολύτως με την καλύτερη διάδοση των εμπειριών αν υπάρχουν ερωτήσεις τις οποίες δεν απάντησα είμαι βέβαιο ότι η Ρεμπέκα Χάρμς θα σας απαντήσει όλες σας τις ερωτήσεις. Ε, εύχομαι ε, στην εισηγήτρια και σε εσά μια πολύ επικοδομητική συνεργασία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καταληκτικά σας σχόλια. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για το σχέδιο έκθεσης είναι η 11η Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. το μεσημέρι. 12 η ώρα το μεσημέρι. Ωραία, τελειώσαμε με αυτό το θέμα και μπορούμε να περάσουμε στο κομμάτι της δημόσιας ακρόασης για τον ορίζοντα Ευρώπη, αριστεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία. This public hearing... Η δημόσια ακρόαση. Παρακαλώ πολύ αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε στις θέσεις σας γιατί η συζήτηση πρέπει να γίνεται ε, μεταξύ όλων και όχι σε πηγαδάκια. Θα ήθελα να προσκαλέσω τους ε, εμπειρογνώμονές μας να καθίσουν εδώ να τους ευχαριστήσω που δέχθηκαν να ε, συμμετάσχουν σημερινή ακρόαση. I have the pleasure. Έχω την χαρά, λέει ο πρόεδρος. Kurt Vandenberg. Να σας παρουσιάσω τον κύριο Κούρτ Βάντενμπεργκ, ο οποίος είναι Διευθυντής του Τμήματος ε, Στρατηγικής Ανάπτυξης και Συντονισμού στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μας κάνει μια παρουσίαση έτσι ώστε να μας ε, ε, κάνει μια σχετική ενημέρωση πριν από την υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού προγράμματος του Ορίζοντος Ευρώπη. Θα μας πει ε, ποιο είναι το περιεχόμενο ε, το, του πιο σημαντικού ε, προγράμματος πλαισίου για την χρηματοδότηση της έρευνας, το Horizon Europe, που υπολογίζουμε να ξεκινήσει την αρχή του 2021. Από τη στιγμή της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης της Κομισιόν την 7η Ιουνίου αρχίσαμε να ε, εργαζόμαστε για το θέμα αυτό ως αρμόδια επί της ουσίας ε, επιτροπής. Επιτροπή. Θέλουμε οπωσδήποτε να υπάρχει και ε, συμφωνία με το Συμβούλιο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Συνειδητοποιούμε βεβαίως ότι είναι δύσκολο να ε, ε, κλείνουν προγράμματα τόσο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κινητοποιηθούμε. Η Επιτροπή Ήτρε είναι όπως είπα η αρμόδια επί της ουσίας ε, για το θέμα αυτό αλλά συνεργάζεται στενά με εννέα επιτροπές οι άλλες οι οποίες θα γνωμοδοτήσουν Envy, Agri, Regi, Cult, Tran προϋπολογισμού, κοντ, ελέγχου του προϋπολογισμού. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να, να καλωσορίσω τους ε, εισηγητές γνωμοδοτήσεων από τις άλλες επιτροπές, την κυρία Κατάινεν επίσης, δεν έχουμε εδώ τον εισηγητή από την Επιτροπή Γεωργίας και να καλωσορίσω και τον Λάμπερτ Βανίστερο, ο οποίος είναι εισηγητή γνωμοδότηση από πλευρά Επιτροπής ε, Περιφερει... Ε, Περιφερειακής Πολιτικής. Α, όχι, δεν είναι ούτε εκείνο εδώ. Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας δυόμιση ώρες. Our rules, we have to finish αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσουμε στις 6 ε, και το απόγευμα. Δεν θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε στις γλώσσες μας παρά μόνο σε αυτή τη lingua franca των Αγγλικών. Μετά από τις 6.30 δηλαδή δεν θα έχουμε δυνατότητα διερμηνίας. Ε, η κάθε παρουσίαση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 10 λεπτά. Παρακαλώ πολύ λοιπόν να είστε ευγενείς και να μην ακολουθήσετε το παράδειγμα των πολιτικών που δεν καταφέρνουν να περιορίσουν τον εαυτό τους στον χρόνο που τους έχει δοθεί. Είμαι υποχρεωμένος ε, να παρακολουθώ στενά τον χρόνο σας και μετά με τις παρουσιάσεις θα δώσουμε το λόγο στους εισηγητές. Λοιπόν, δίνω το λόγο αμέσως στον κύριο Βάντενμπεργκ, ο οποίος θα κάνει την εισαγωγή για το όλο θέμα. Κύριε Βάντερμπεργκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να κάνω κάποιε εισαγωγικέ παρατηρήσει σε αυτή την ακρόαση. Είναι ευγνώμων η Κομισιόν στο Κοινοβούλιο αλλά και στην Ήτρε που οργάνωσε αυτή την ακρόαση όλων των ενδιαφερομένων μερών. Πρόθεσή μα ήταν να παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μία πρόταση που θα μπορούσε να κινητοποιήσει του πάντε που θα μπορούσε να κινητοποιήσει οργανισμούς, ανθρώπους και ε, ακόμα περισσότερο. Χαιρόμαστε που ο Horizon Europe είχε ήδη αυτήν την ε, δύναμη κινητοποίησης και που ξεκίνησε τόσο γρήγορα η σε βάθος ε, μελέτη της πρότασης ε, με όλους τους εισηγητές και συνεισηγητές. Ε, ξέρουμε ότι έχουν μελετηθεί 4.000 τροπολογίες ε, είναι πολύ εμπλεκόμενοι, τους ανέφερε εν μέρη ο Πρόεδρος. Ε, χαιρόμαστε ότι δεν έχει λησμονηθεί και η πρόταση ε, Euratom και ευχαριστώ την σχετική εισηγήτρια. Βλέπουμε ότι και από πλευράς του Συμβουλίου τα πράγματα έχουν επιταχυνθεί ε, Στην 28η Σεπτεμβρίου στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού ακούσαμε από τα χείλη των Υπουργών ότι όλοι κινητοποιούνται με γοργό ρυθμό. Η κινητοποίηση αυτή ε, λαμβάνει η χώρα και μεταξύ των υπουργων οτι ολοι κινητοποιουνται με γοργο ρυθμο η κινητοποιηση αυτη λαμβανει χωρα και μεταξυ των εμπλεκομενων και των ενδιαφέρων μερών. Έχουμε ε, πολλές επιστροφές και ανταποκρίσεις όσον αφορά τις πλήστες δημόσιες διαβουλεύσεις που έχουν λάβει χώρα και πιστεύουμε ότι πραγματικά το πρόγραμμα ε, πλαίσιο θα έχει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία από τη σήμερα στο μέλλον. Η Κομισιόν συμφωνεί με το κεντρικό θέμα του της ακρόασης πώς ε, θα πρέπει να, να, να ε, προχωρήσει το πρόγραμμα Horizon Europe έτσι ώστε να αποδώσει τα μέγιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην έρευνα και την καινοτομία. Είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι επί της ουσίας ε, να αναλάβουν την ιδιοκτησία του προγράμματος γιατί από αυτούς εξαρτάται και προωθείται η ε, επιτυχία. Ε, μιλάμε βέβαια και για τις επιχειρήσεις μικρές και μεσές ή και μεγαλύτερες και επομένως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ανοίξουμε το πρόγραμμα όσο γίνεται σε περισσότερο κόσμο και σε νεοαφιχθέντες αλλά και νέους φορείς όπως είναι ας πούμε οι δημοί οι κοινότητες. Εμείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέλαμε ε, ε, συνδημιουργία ε, και αυτή η συνδημιουργία να αποτελέσει το βασικό, το βασικό στοιχείο του DNA, το βασικό χαρακτηριστικό λοιπόν αυτού του προγράμματος. Θέλουμε να οργανώσουμε αυτήν την συνδημιουργία έτσι ώστε η ευρωπαϊκή υλοποίηση να μην αποτελεί μια σειρά κάλυψης ενδιαφερόντων μεμονωμένων ενδιαφερομένων ή εμπλεκομένων, αλλά θέλουμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι από κοινού ε, να ε, εργαστούν. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μονάχα να αναρωτηθεί κανείς τι μπορεί να δώσει αυτό το πρόγραμμα σε μένα, αλλά τι μπορεί να δώσει στο σύνολο της Ευρώπης το πρόγραμμα αυτό. Horizon Europe. Ε, είναι ε, γεγονός ότι πρέπει να μάθουμε τα μαθήματα που μας δίδαξε το ορίζοντας 2020 ε, και να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία στρατηγικού σχεδιασμού, θα αναφερθώ αργότερα σε αυτά, αλλά τρεις στόχους που θα καλυφθούν και από τις παρεμβάσεις σήμερα ο πρώτος στόχος είναι η μεγιστοποίηση του αντικτύπου στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού ε, πρέπει να είναι να δώσει ένα πραγματικά στρατηγικό εργαλείο για τον τρόπο με τον οποίο ε, μπορεί, μπορούμε να έχουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο ε, ανάμεσα από τον συνδυασμένο κύκλο ενεργειών για την έρευνα και την καινοτομία. Δεν μας ενδιαφέρουν με μονο, μια μυριάδα, ας πούμε, μια πληθώρα μεμονωμένων εργαλείων. Θέλουμε με στρατηγικό σχεδιασμό έτσι ώστε η υλοποίηση του προγράμματος να, να ε, ε, ταυτίζεται με την διαρκώς ε, με την κατάσταση που διαρκώς αλλάζει, με την διαρκώς εναλλασσόμενη κατάσταση όσον αφορά και τις προκλήσεις ε, και τις ε, γνώσεις. Θέλουμε επίσης ε, καλή ισορροπία μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας. Θέλουμε επίσης να υπογραμμίσουμε το ρόλο της κοινωνίας μέσα σε όλα αυτά. Τον ρόλο της διαλειτουργικότητας, τον ρόλο της, του, του φύλου, την διάσταση μάλλον του φίλου την διάσταση της ισότητας όσον αφορά ε, όλο ε, αυτό το εγχείρημα και φυσικά ε, και τον ρόλο της δια Δεύτερο στοιχείο, πολύ σημαντικό, είναι η διαφάνεια αυτό θα είναι καλό για όλους τους εμπλεκόμενους. Στον ορίζοντα 2020 ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορούσε μια εσωτερική διαδικασία και υπήρχαν μονάχα κάποια έγγραφα τα οποία ήταν ανοιχτά ε, και ε, δημοσιοποιημένα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός τώρα του νέου προγράμματος ε, θέλουμε να μας δώσει την δυνατότητα της δημιουργίας ενός ενίου εγγράφου που θα αναφέρει τους στόχους της Κομισιόν πριν από το σχεδιασμό των μεμονωμένων προγραμμάτων όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι προτάσεις και θέλουμε βεβαίως και feedback, ανάδραση από τους ενδιαφερόμενους που είτε θα ακυρώσουν είτε θα επικυρώσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό πριν γίνει guiding document. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει πραγματικά συνδημιουργία. Οδηγούμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό στον τρίτο στόχο Θέλουμε στρατηγικό σχεδιασμό που να μπορεί να δημιουργήσει ένα θεματολόγιο αναφοράς για τα, προγράμματα, για τα εθνικά προγράμματα ε, έρευνας και ε, καινοτομίας ε, και με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσουμε συνέργειες ή να διευκολύνουμε τις συνέργειες μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων πάντα έχοντας ε, το βλέμμα από άποψη στρατηγικής στραμμένο προς το στρατηγικό σχεδιασμό του ορίζοντα Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει λοιπόν και η σχέση ανάμεσα στο Horizon Europe ε, από τη μία πλευρά και τα περιφερειακά προγράμματα, τα ε, ταμεία, τα διορθωτικά ταμεία κλπ. Η Κομισιόν προτείνει έναν αποτελεσματικό, συνολικό και διαφανή ε, ε, ε, τρόπο εργασίας για τον στρατηγικό σχεδιασμό που όμως δεν βαραίνει γραφειοκρατικά την όλη διαδικασία και ευελπιστούμε ότι θα γίνει καλοδεχούμενος ο στρατηγικός αυτός σχεδιασμός από όλους. Νομίζω ότι όλοι θέλουν ε, σαφήνεια και ε, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας την 28η Σεπτεμβρίου ακούσαμε τις απόψεις και των κρατών ε, μελών που θέλουν να ακολουθήσουν την δυτή πορεία που προτείνει η Αυστριακή Προεδρία. Δηλαδή συνεργασία όσον αφορά την ε, νομική ε, βάση ε, και για τα υπόλοιπα εκτελεστικές πράξεις. Ξέρετε ότι θα υπάρξει και ένα επίσημο γεύμα που θα αποτελέσει με της συζήτησης σχετικά με το τι θα μπορούσαν να είναι οι θεσμικές εταιρικές σχέσεις, institutional partnerships, είναι πολύ σημαντικό να ε, διατηρηθεί το θέμα αυτό σε, ε, ε, σε περιοχές έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αλλάζει η νομική βάση και να ευθυγραμμιστεί και με την αρχική ιδέα που είχαμε όσον αφορά το, την συναντήληψη και την συνδημιουργία. Επίσης έχουμε συμφωνήσει ότι θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη με ταχύ ρυθμό σχετικά με το πώς θα είναι το, ο υπόλοιπος στρατηγικός σχεδιασμός και το θεσμικό πλαίσιο. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι μέλη του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε ε, να συγχαρεί το Κοινοβούλιο για την διαρκή υποστήριξη ε, και στα πλαίσια του προϋπολογισμού για το 2019, διότι το Κοινοβούλιο πιέζει έτσι ώστε ε, να ε, επαναδιατυπωθεί ο προϋπολογισμός έτσι όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Για μας είναι πολύ πιο εύκολο βεβαίως να διαχειριστούμε περισσότερους παρά λιγότερους πόρους. Χαιρόμαστε που και στον ορίζοντα 20 υπάρχει μεγάλη ε, ε, ορμή ε, κατά την συζήτηση. να είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να λυθούν ε, ε, αλλά είναι γεγονός ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες οι οποίες δεν είναι αυτονόητες για τη συμπερίληψη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Είμαστε ωστόσο πεπισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν ε, βλέπουμε ισχυρή αμφισβήτηση όσον αφορά την κεντρική στόχευση του Horizon Europe. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο και γι' αυτό λοιπόν τώρα θα ήθελα να ακούσω από τους εμπλεκόμενους πώς βλέπουν το Horizon Europe και πώς μπορούν να συμβάλλουν στην πλήρη επιτυχία Το Ευχαριστώ. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, ε, ξεπεράσατε 10% των χρόνων που σας είχαμε δώσει. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις συζητήσεις μας και θα τις σε δύο τμήματα. Καταρχάς, θα γίνει μία παρουσίαση από τον καθηγητή Σεντόσκη και μετά από την κυρία Σαμπίνες Λέσκα. Το λόγο έχει ο κύριος Παλμόφσκι. Συμφωνείτε? Μάλιστα. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ήτρε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για την πρόσκλησή σας, αλλά και για την υποστήριξή σας, ε, την τερκή υποστήριξή σας στην έρευνα και στην ανάπτυξη ενός πιο φιλόδοξου προγράμματος για το Horizon Europe. Εκπροσωπώ την ε, Ένωση 19 κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων συμπεριλαμβανομένων και των 15 κρατών μελών. Το βασικό μου μήνυμα είναι ότι το Horizon Europe θα εκπληρώσει το δυναμικό του αν υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ Έρευνα και καινοτομία. γιατί θεωρούμε ότι επικεντρώνεται το πρόγραμμα της ε, ε, Επιτροπής υπερβολικά πολύ στην καινοτομία εις βάρος τη επιστήμης. Να μιλήσω για τη σημασία της ε, επιστημονικής αριστείας. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο του Horizon Europe και είναι το σημείο κίνησή μου, γιατί είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία του Horizon. Κανένα κράτο μέλο όσα και ένα δαπανά στην έρευνα δεν μπορεί να πατύχει το αποτέλεσμα αυτό, γιατί ο Horizon είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει τις, ε, τα προγράμματα αυτά διασυνοριακά. Είναι κάτι μοναδικό πραγματικά και γι' αυτό λοιπόν το πρόγραμμα Horizon ε, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους τους επιστήμονες παγκόσμια. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όμως, γιατί η φήμη είναι κάτι το οποίο παίρνει πολύ χρόνο να δημιουργηθεί και καταστράφεται πολύ γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, μετατόπιση των συνόρων. Ναι. Επίσης, ε, θα πρέπει να συστήνονται ομάδες ε, συμβουλευτικές για να υποστηρίζουν. Άρα, θα πρέπει να φροντίσουμε ότι το Horizon Europe θα υποστηρίζει την αριστεία. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην κλείσουμε το χάσμα μεταξύ των 15 και των 27. Γιατί αυτός ο στόχος θα υπονόμευε τους στόχους του ορίζοντα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μας απασχολεί το κενό αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αυξηθεί από 1,8% στο 2,5% για την, το Sharing Excellence. Επίσης, την ε, τυφλή αξιολόγηση των ε, προτάσεων. Δεν ε, βλέπουμε γιατί να μην ισχύσει κάτι τέτοιο για το Horizon 2020. Και τέλος, να υπάρχει ποικιλία των ερευνητών σε τεφαρά το φύλλο, την περιοχή, αλλά ποτέ αυτό εις βάρος της αριστείας. Να είναι μόνο μία αρχή όταν είναι ίσως οι προτάσεις. Επίσης, το πρόγραμμα Sharing Excellence θα πρέπει να ισχύει για περιφέρειες, όχι μόνο για χώρες. Επίσης, αμφιβάλλουμε για το κατά πόσο έχει νομική βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα βασικό θέμα, λοιπόν, είναι η ανησυχία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί παγκόσμια ηγέτη σε ό,τι αφορά την έρευνα, αλλά δεν έχει αντίστοιχη θέση σε ό,τι αφορά την κοινοτομία. Οι δράσεις Μαρίς Κλεντόφσκα Κιουρί θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν, αλλά για τον πυλώνα 2 και 3 επικεντρώνονται σε θέματα που είναι σχετικά με την αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει το μεριδιό τη και την ε, πρώτη καθηγητρία τη σε ό,τι αφορά την παραγωγή επιστημόνων λόγω τη Κίνα από 3 από το 17% λοιπόν το 2017. Είναι μεγάλες οι απώλειες και είναι και σκληρός ο αγώνας. Γι' αυτό λοιπόν το... η υποστήριξη των νέων επιστημόνων θα πρέπει να συνεχιστεί παρατέρων. Λοιπόν, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Στέφαν Παλεσκή προβλέπονται σχετικά βραβεία τα οποία οδηγούν σε βραβεία Νόμπελ. Ο Μπεν Φούριγκερ, διάδοχος ε, νομπελίστα στη χημεία το 2016 και αυτός ήταν προμευμένος από το MSCI. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν το ίδιο πράγμα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομίες στα νέα ταλέντα μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε από τις πιο επιτυχείς οργανώσεις σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των κορυφαίων ε, ερευνητών. Αλλά σήμερα μόνο το 20% των προγραμμάτων χρηματοδοτείται λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, έλλειψη πόρων. Είναι τεράστιες ε, οι απώλειες που προκαλούνται έτσι. Θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικό λοιπόν τα κονδύλια αυτά και επίσης και τη συνεργατική επιστήμη θα πρέπει να ενισχύσουμε. Οι σχετικές ε, ευκαιρίες στο Horizon 2020 λείπουν γιατί κοιτάμε πιο πολλές λύσεις ε, που μπορούν να εμπορευτούν. Και αυτό μετά, αυτό συνεχίζεται μάλλον και στο Horizon Europe. Τα πανεπιστήμια όλα ζητούν να υποστηριχθούν και να βοηθηθούν σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ ότι επικεντρώνονται μαζικά στις νέες τεχνολογίες. Χρειαζόμαστε νέες τεχνολογίες, φυσικά και τις χρειαζόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, να μην ξεχνάμε όμως τους ε, βιώσιμού στόχους της χιλιετίας. Ανησυχούμε, ανησυχούμε για την παγκοσμιοποίηση, τη μετανάστευση, την εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό απασχολεί τον πολίτη και αυτό εκφράζεται και στις εκλογές. Άρα θα πρέπει να επενδύσουμε σε τέτοιου είδου προκλήσεις, σε τέτοιου είδου προσκλήσεις. Να μην επικεντρωθούμε λοιπόν μόνο στην τεχνολογία. Πολύ καλή είναι η τεχνολογία, αλλά υπάρχουν και άλλες προκλήσεις σε κοινωνικό επίπεδο για να, λάβουμε, για να πάρουμε στα σοβαρά τις ανησυχίες του πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στις τεχνολογικές λύσεις, αλλά στις ανάγκες τη κοινωνία, νέου τρόπους για να αλλάξουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο και αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω επιστημονικής καινοτομία. και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται και στη χρηματοδότηση. Όταν μιλάμε για τις κοινωνικές ανάγκες της Ευρώπης, κοινωνικές επιστήμες, σημαντική χρηματοδότηση αυτών, το Horizon 2020 έχει τόσο χαμηλή ποσοστό επενδύσεων που είχαμε μόνο ένα ποσοστό επιτυχίας 4,4%. Είναι μεγάλη λοιπόν η έλλειψη τέτοιων προγραμμάτων. Θα πρέπει να πετύχουμε κάτι καλύτερο για το Horizon Europe. Θα πρέπει να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για τέτοια κοινωνικά θέματα. Είναι επίση κρίσιμο να υπάρξει ένταξη και να αποτελέσει αυτό στρατηγικό στόχο του προγράμματος. Δεν μπορούμε να το αντικαταθίσουμε αυτό με κάποιες υποσχέσεις για εγκάρσια ένταξη των θεμάτων αυτών. Θα πρέπει να υπάρχει η ένταξη των θεμάτων αυτών ε, στο Horizon ε, Europe. Και τέλος, δεν ε, μπορεί να αντικατασταθεί από άλλα προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το πρόγραμμα Creative Europe. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις αλληλεπικαλύψεις. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια συμμετοχική κοινωνία και να μην υπάρχει διπλή χρηματοδότηση. Τέλος, Τι ημέρε αυτέ ακούμε πολύ συχνά ότι θα πρέπει να μπουν τα συμφέροντα τη Ένωση πρώτα. Η μοναδική όμως προστιθέμενη αξία του Horizon Europe είναι η συνεργασία των καλύτερων μυαλών υπέρ του συμφέροντο της Ευρώπης. Το να βάλουμε λοιπόν την ευρωπαϊκή τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα πρώτο και πάνω απ' όλα. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό συνεργασίας εδώ. Αυτό το ποσοστό λοιπόν ένταξη θα πρέπει να αυξηθεί. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως ε, φυσικά βάσει και των ε, συμφωνιών ε, προσχώρησης. Κυρίες και κύριοι, να συνοψίσω με τα πέντε αυτά σημεία τα οποία τα βλέπετε και στη διαφάνεια. Καταρχάς, να σας πω ότι σήμερα το Horizon Europe δεν έχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης βασικής έρευνας ε, της επιστήμης και καινοτομία. Και αν δεν καταφέρουμε να συνδέσουμε το πρόγραμμα με τους βιώσιμους στόχους, δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε την, ε, τις απαντήσεις ε, στα βασικά κοινωνικά προβλήματα και δεν έχουμε τίποτε στο οποίο θα θέλουμε να καινοτομήσουμε. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε γενικά την ευρωπαϊκή επιστήμη και το Horizon Europe μας δίνει μια ευκαιρία να το κάνουμε αυτό, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους ε, επιστήμονες, αλλά για το μέλλον της Ευρώπης και της ε, κοινωνίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και το χρονικό όριο. Από χρονική απόψεω ε, ήσασταν άψογο επίση. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην δόκτωρα Σαμπίν Χελίτσκα. Θα μιλήσω αγγλικά. Έχω μια παρουσίαση. Κυρία, ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά ε, μέλη της Επιτροπής, ε, είναι μια τεράστια ευκαιρία για μας. Εγώ προέρχομαι από την Αυστρία. Ε, η, η Infineon είναι μια εταιρεία ημιαγωγών ε, 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση σε έναν ε, νέο, νέας τεχνολογίας ε, τομέα ε, κατασκευής chip στην Ευρώπη. Είναι μια τεράστια επένδυση, μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή σε αυτό το τομέα στην Ευρώπη. Εμείς πιστεύουμε στην Ευρώπη, επενδύουμε σε αυτήν και δημιουργούμε αγορές, ε, καταστήματα στην Ευρώπη. Βλέπετε εδώ τα σημεία που θα ήθελα να καλύψω θα ήθελα να ξεκινήσω με το να θέσω ε, το πλαίσιο, δηλαδή τι θέλουμε να επιτύχουμε. Καταρχάς υπάρχουν ε, οι μεγάλες τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπετε εδώ μερικές από τις σημαντικότερες. Τις γνωρίζετε όλες, ε, Είναι προκλήσεις, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι είναι και τεράστιες ευκαιρίες για μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα το ζήτημα το ενεργειακό έχετε, ε, το, λό, έχετε το όριο του, της αύξησης θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό. Ε, αυτό είναι τεράστια πρόκληση για μας. Η ψηφιοποίηση είναι επίσης μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη. Ένα θέμα λοιπόν είναι το θέμα του να θέσουμε το πλαίσιο μας. Το δεύτερο είναι τι συμβαίνει γύρω μας. Η Ευρώπη είναι και μπορεί να είναι ένας παγκόσμιος παίκτη πολύ σημαντικός αναφέρθηκε η Κίνα ε, εγώ δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες παρόλο που αναφέρω την Κίνα ευχαρίστως ε, να το κάνω κατά ε, τη συζήτηση μετά αλλά θα ήθελα να πω για τη στρατηγική Made in China 2025 οι Κινέζοι τονίζουν τα σημαντικότερα σημεία το δεύτερο όμως η δεύτερη πτυχή του τι συμβαίνει συμβαίνει γύρω μας και θα σα δώσω και μία παρά, ένα παράδειγμα η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πάρα πολύ σαφείς ως προς την ταχεία ε, ενίσχυση, την ταχεία ε, προώθηση τη τεχνητή νοημοσύνης δείτε εμεί ω Ευρώπη που είμαστε σε αυτό το διάγραμμα ε, το τεράστιο δυναμικό που υπάρχει πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη εκτιμάται εδώ και πάλι χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες βλέπετε στη διαφάνεια βλέπουμε όμως ότι μιλάμε για επίπεδο τρισεκατομμυρίων ε, κάτι ακόμη ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για μας είναι το εξής, ότι όλα αυτά δεν αφορούν μόνο την τεχνολογία. Ε, στην ουσία είμαστε σε μια κοινωνική, πολιτική και οικονομική, σε έναν οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό ανταγωνισμό για τις βασικές μας αξίες και αυτός ο ανταγωνισμός σήμερα ε, αποφασίζεται από την επιστήμη, ε, την έρευνα και την τεχνολογία. Βλέπετε εδώ πλατφόρμες που θεωρούνται το νέο πετρέλαιο. Η Ευρώπη έχει 4% μερίδιο των ε, παγκοσμίων ε, πληροφοριών ε, πλατφορμών δεδομένων. Ήταν εδώ ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ ε, στη συζήτηση μαζί του μπορεί να είχατε την εντύπωση ότι δεν καταλάβαινε πολύ καλά ποιο είναι το ζήτημα ε, όσον αφορά την ε, επεξεργασία των, της ιδιωτικότητας των δεδομένων ή των δεδομένων στην, κοινό στην Κίνα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα που απλώς εφαρμόζει τις αξίες της κοινωνίας τους. Ε, η τεχνολογία λοιπόν υπάρχει περίπτωση να ε, επηρεάσει τις κοινωνικές μας ανάγκες, την αυτονομία μας και την κυριαρχία μας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν ε, είναι επιστημονική φαντασία, είναι κάτι που συμβαίνει στο περιβάλλον μας θα ε, έρθω τώρα σε αυτό που πρέπει να ε, πραγματευτώ για σήμερα ε, όσον αφορά τις συμπράξεις. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, συμπράξεις δημοτικού και, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τα σχετικά προγράμματα. Θα ήθελα να περάσω κατευθείαν στην ουσία πάντοτε υπάρχει προστιθέμενη αξία και αντίκτυπος των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και αυτό μπορεί να συνοψιστεί καλύτερα επειδή δημιουργεί μια κρίσιμη μάζα, ε, συγκεντρώνει τις ιδέες, ε, τις απόψεις, ε, των τις επενδύσεις, καταλήγουμε σε ένα μακρο, μακροπρόθεσμο όραμα και έτσι ενισχύουμε το ευρωπαϊκό οικοσύστημα σε συνεργασία με την επιστήμη, με την έρευνα και την τεχνολογία και όλους τους εταίρους του οικοσυστήματός μας. Εμείς ε, δίνουμε το δικό μας μερίδιο στην οικοδόμηση αυτής της κοινή Ευρώπης. Όσον αφορά το Excel, επειδή μου ζητήθηκε να ε, το ε, σχολιάσω, ειδικότερα τις ηλεκτρικές συνιστώσεις, εμείς ενισχύουμε και, και την ψηφιοποίηση, το αναλογικό και το ψηφιακό τα συνδέουμε για να μπορέσουμε να επιφέρουμε την ψηφιοποίηση, να την καταστήσουμε δυνατή και κάνοντας το αυτό και οι ιδιώτες και οι δημόσιοι φορείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη συνεργάζονται και αυτό δημιουργεί μια τεράστια προστιθέμενη αξία, όπω βλέπετε εδώ από τα αριθμητικά στοιχεία. Το δυναμικό για την Ευρώπη είναι και πάλι τεράστιο βάσει των ε, ηλεκτρονικών συνιστοσών και των συστημάτων. 50% ε, του ευρωπαϊκού ΑΕΠ μέχρι το 2020 ε, βασίζεται στις στα, στα ηλεκτρονικά συστήματα και τις συνιστώσεις τους. Στην ουσία δηλαδή αυτές ε, οι κοινέ ε, συμπράξεις, ε, βλέπετε εδώ μερικά στοιχεία, βλέπετε τι αφορούν, έχουν, είναι, έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή, αφορούν την επιστολή όχι το μέσο και επίσης αφορούν και τον αντίκτυπο. Έχουν χρηματοδότηση και είναι αποτελεσματική και ως προς το κόστος. Για παράδειγμα στο Excel βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τριμερές μοντέλο με τρία σκέλη για να το πω καλύτερα και υπάρχουν, πρέπει να δημιουργήσουμε τις τεχνολογικές ε, ικανότητες τις απαραίτητες για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την τεχνολογική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι χρειάζεται τώρα για το μέλλον σε σχέση με ε, τις κοινοπραξίες αυτές. Αυτό που ε, ζητούμε είναι να υπάρξει μια συνειδητοποίηση του στρατηγικού και πολιτικού ρόλου των ε, κοινοπραξιών αυτών και να υπάρξει και μεγάλη επένδυση από πλευράς, μάλλον στους τομείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, ε, οι ιδιωτικοί φορείς. Ε, αυτό αποτελεί έναν πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα που μπορεί να βοηθήσει στον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο της επένδυσης. Όλα τα μέτρα χρειάζονται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το επίπεδο, το περιβάλλον χαμηλής ανταγωνιστικότητας που ανέφερα προηγουμένως. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη εμβέλεια, χρειάζεται υψηλότερο προπολογισμό που θα συνάδει βέβαια με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και υπάρχουν και κάποια ζητήματα με τις προϋποθέσεις ε, για να υπάρξει για παράδειγμα ε, καλύτερη χρηματοδότηση και καλύτερη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων. Και θα ήθελα ολοκληρώνοντα να τονίσω ότι ε, το νέο γεωπολιτικό νόμισμα είναι η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία και συνεπώς ε, η οικονομική αυτονομία, η κυριαρχία και η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικά για το περιβάλλον μας. Χρειαζόμαστε την αίσθηση του κατεπήγοντος σε σχέση με τα τολμηρά ε, μέτρα ε, και όσον αφορά τη στρατηγική και όσον αφορά την επένδυση και όσον αφορά την ταχύτητα. Και οι κοινοπραξίες είναι σημαντικά μέσα με πραγματική προστιθέμενη αξία και απτά αποτελέσματα. Αυτό έχει αποδειχθεί θα μπορούσα να το εξηγήσω και διαφορετικά. Βάσει όλων όσων κατέδειξα ε, θα έπρεπε να πω ότι η, ε, ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη και περισσότερες από τις βασικές μας αξίες και εμείς οι, οι, οι κοινοπραξίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ε, οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε πιο επιτυχείς, να ε, προχωρήσουμε, να αυξήσουμε το μερίδιό μας παγκοσμίω και να αυξήσουμε και την ανταγωνιστικότητά μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω την δέσμευσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. χρονικός, ήσασταν επίσης άψογοι. Λοιπόν, Επόμενος ομιλητής, μάλλον θα έχουμε εισαγωγικές παρατηρήσεις από δύο εισηγητές μας. Να ζητήσω λοιπόν τον κύριο Ντανίκα πρώτα να ξεκινήσει με τις πρώτες του παρατηρήσεις. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά αγαπητοί συνάδελφε και μετά ο κύριος Σάρεπα αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ So, uh, in, uh, in preparing this report, uh, I, I had the chance to, to meet some of you. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω μερικούς ε, ε, από εσά και χαίρομαι, και χαίρομαι που είσαστε εδώ και μπορούμε να συζητήσουμε. Θα ήθελα όμως ε, να συζητήσουμε κάποια ζητήματα και να αναφέρω εγώ μερικά. Πιστεύουμε ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για το Horizon Europe. Η Κομισιόν νομίζω δεν ξέρει. Εσείς βέβαια τα ξέρετε και από πρώτο χέρι γιατί δουλεύετε με τις επιχειρήσεις ή δουλεύετε με την έρευνα. Αλλά τι, ποια είναι η θέση του Ευρωπαίου πολίτη. Γιατί αυτοί πληρώνουν τελικά τους φόρους. Αυτοί είναι οι φορολογούμενοι. Και κάπου χάνουμε τη θέση του Ευρωπαίου πολίτη που λέει «ΟΚ, να πληρώσω τους φόρους μου, αλλά ποια θα είναι η επιστροφή των χρημάτων ε, που έχω πληρώσει» θα ήθελα βεβαίως να καλωσορίσω ε, την ε, αρχή της Guild που ανέφερε ο κύριος Παλμόφς και προηγουμένως Europe First, πρώτα η Ευρώπη. Αλλά δεν έχουμε και τόσα χρήματα για να τα μοιράζουμε σε όλο τον κόσμο. Ε, και τρεις από, τις, ε, από κάθε τέσσερις εξαιρετικές προτάσεις ε, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Γι' αυτό λοιπόν το Europe First και όσον αφορά τη θέση της Κομισιόν και όσον αφορά ε, την υποστήριξη των προγραμμάτων. Ε, πρέπει σε όλα αυτά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αντιαποτελεσματικοί. Απ' την άλλη μεριά λέμε ότι ε, πρέπει να υπάρχει σωστός ανταγωνισμός. Ναι, οπωσδήποτε. Αλλά ε, οπωσδήποτε θα πρέπει ε, αυτό να φαίνεται καθαρά. Ε, ο κύριος Βάντενμπεργκ μας είπε ότι συζητήθηκε το θέμα στους στα πλαίσια του Συμβουλίου των Υπουργών και ένας ε, υπουργός ε, είπε ότι θα πρέπει να μελετώνται καλά τα, τα προγράμματα ε, και Μάλιστα ένας υπουργός είπε ότι υπήρξε ένα πρόγραμμα που αξιολογήθηκε θετικά από που το έτρεχε μάλιστα ένας μελετητής που είχε κερδίσει βραβείο Νόμπελ και απέτυχε, απέτυχε ε, το πρόγραμμα αυτό και ε, ε, και τελικά η Κομισιόν είπε ναι δεν έγινε σωστή αξιολόγηση και μετά όταν συζητήθηκε το θέμα με τον επιστήμονα που είχε κερδίσει τον Νόμπελ είπε ότι χαίρομαι που δεν έγινε ξέρετε ήταν μια ιδέα ανόητη του βοηθού μου και εν πάση περιπτώσει δεν έγινε σωστή η αξιολόγηση. Πιστεύω ότι ε, ε, πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, θα πρέπει να δαπανίσουμε τα χρήματα ε, με τρόπο ώστε πραγματικά να ωφεληθούν οι πολίτες της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. You can see uh, the Βλέπετε βέβαια και την διαφορά ανάμεσα στους ε, πολιτικούς ε, και τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες ζητούν ένα 10% ε, ενώ οι πολιτικοί ζητάνε 30% και παραπάνω 100%. Επόμενος συνάδελφος παρακαλώ. Φυσικά δεν μπορώ να συμφωνήσω Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την ιδέα ότι οι δύο ε, οι ε, οι οποίοι αναφέρονται σε ένα πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ ε, και που μπορούν να επηρεάσουν τη θέση του Κοινοβουλίου να έχουν τρία λεπτά να μιλήσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Με τον στρατηγικό σχεδιασμό μπαίνουμε σε μια ιδιάζουσα κατάσταση. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο έχει η αρμοδιότητα ε, να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει ασφάλεια ε, στους ε, επενδυτές και ε, τεχνογνωσία, σωστή χρήση της τεχνογνωσίας. Δεν ξέρω αν με συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού ή χωρίς, πάντως οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε έναν σωστό σχεδιασμό. Το Κοινοβούλιο έχει υποβάλει κάποιες προτάσεις μέσω των οποίων εκφράζει την ε, εμπιστοσύνη του στην Κομισιόν. Το ζήτημα πάντως είναι ε, να προχωρήσουμε την υλοποίηση όσο γίνεται περισσότερο και όσο γίνεται πιο μακριά. Ίσως θα μπορούσα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις και να τις απαντήσετε αργότερα. Σε σχέση με τεχνολογία IT, ίσως ε, μπορεί να έχουμε κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε ορισμένους τομείς. Ίσως να έχουμε ε, ένα προβάδισμα ενός ενάμιση έτους σε ορισμένους ε, τομείς. Ωστόσο, μέχρι ποιο βαθμό πιστεύετε ότι είναι πιθανό στις διαπραγματεύσεις για να δημιουργήσουμε αυτά τα ευραία κονσόρσιου, αυτές τις συμπράξεις τις ε, ευρείες ε, εάν δεν μπορεί να ακολουθήσει και ο προϋπολογισμός γιατί θα πρέπει να δούμε μέχρι ποιο βαθμό είμαστε σε, είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε τέτοιες συμπράξεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Επίσης, ε, καλά τα λέτε κύριε Παλμόφσκι, αλλά μην το παρακάνετε και με το Κοινοβούλιο το κοινοβούλιο λέτε αύξησε το προϋπολογισμό, ναι, αλλά ε, εάν ε, ε, έρχεστε εδώ και κάνετε σαν ανταγωνισμό ανάμεσα σε εσά και τους άλλους και κάποιους άλλους ε, δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ζήτημα είναι να έχουμε ένα, μια ισχυρή φωνή με την οποία θα μιλήσουμε όλοι μαζί και δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ε, διαχωρισμός ε, του προγράμματος ε, στα δύο όπου το ένα θα είναι οι ανάγκες της κοινωνίας και το άλλο θα καλύπτει οι άλλες ανάγκες. Το ζήτημα είναι αν μπορούν να υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε, να υλοποιήσουμε τα προγράμματα αυτά. Επίσης, στην ουσία όλοι οι αύξησαν τον, τον προϋπολογισμό και πιστεύω ότι δεν είναι το πρόβλημα το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να πάτε στα κράτη-μέλη και να συζητήσετε γιατί το θέμα δεν είναι αν μας αρέσει ή όχι αυτό το SSH που αναφέρατε εσείς, αλλά τα χρήματα τα οποία μπορούν να υπάρχουν ε, και είναι γεγονός ότι ε, εδώ μιλάμε για αποφάσεις που έχουν πάρει τα κράτη-μέλη ε, τα οποία δεν έχουν αποφασίσει να δώσουν χρήματα για το SSH. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Dank. Δεν εξαντλήσατε και το χρονικό όριο που σας είχαμε δώσει. Να περάσουμε στους κοιόδης. Ο πρώτος ήταν ο κύριος μάλλον. Από το ΕΛΚΑ. Κάμπεθό νωρίς. Από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Είναι η δεύτερη. Madame ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, παρεμβαίνοντες ε, να, υποστηρί... να υπογραμμίσω για κάποια στοιχεία και να κάνω και κάποιες ε, ερωτήσεις. Βεβαίως το μέλλον θα είναι ψηφιακό, θα είναι τεχνολογικό, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ε, και τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και να διασυνδέσουμε την επιστήμη με αυτές τις αξίες. Η η επιστήμη μπορεί να είναι όχημα και πιστεύω ότι αυτό το επίκεντρο των ε, αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηριχτεί είτε σε απλές επενδύσεις είτε σε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Εν πάση περιπτώσει αυτό που είναι σημαντικό είναι το τελικό αποτέλεσμα να φτάσει στους ε, πολίτες. Αριστεία. Χρειαζόμαστε περισσότερη αριστεία. Χρειαζόμαστε περισσότερες περιφέρειες που θα έχουν την αριστεία αυτή. Θα πρέπει να διευρύνουμε επεκτείνουμε την ε, ικανότητα αυτή για αριστεία. Θα πρέπει να ευημερήσει κατά κάποιο τρόπο αυτή η αριστεία. Και οπωσδήποτε ε, στα πλαίσια αυτής της αριστείας θα πρέπει να βρουν τη θέση τους και να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι περιφέρειες ε, τις οποίες πρέπει να υποστηρίξουμε. Να υποστηρίξουμε επίσης και τους νέους. Οι νέοι οπωσδήποτε θα πρέπει να αποκτήσουν, να ενσωματωθούν σε αυτήν την ε, διαδικασία και υπάρχουν ε, ταλέντα τα οποία λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν σιωπήσει. Θα πρέπει αυτό να σταματήσει. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Είναι το, η πρόταση της ε, ε Κομισιόν δεν το συμπεριλαμβάνει και δεν το αντιμετωπίζει σωστά. Είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ε μπορούν, πρέπει να έχουν και οι μικρές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτές τις δομές. Όχι μονάχα οι μεγάλες άλλες ε, μονάδες. Επίσης, ε, ο επιχειρηματικός ε, μη χρηματοπιστωτικός τομέας θα πρέπει να υποστηριχθεί. Και να πούμε ότι οι περισσότερες από το 23% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν απασχολούν λιγότερο από 10 άτομα προσωπικό και αυτές συνήθως μένουν απ' έξω. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το εργαλείο αυτό σωστά ε, και ε, να έχει, μεγάλη, ε, έχει μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για κάθε ευρώ μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορούμε να έχουμε επιστροφή 1,6. Και μία τελευταία ερώτηση. Όταν Μιλάμε ε, για ένα εργαλείο ειδικού σκοπού ε, που θα διαχειριστεί το δημόσιο χρήμα. Δεν μπορώ να πω ότι αντιτίθεμαι, αλλά ε, γιατί θέλουμε αυτό το, δημόσιο χρήμα να το αντιμετωπίσουμε με ειδικό τρόπο. Ευχαριστώ. και εσείς χρησιμοποιήσατε σχεδόν το 100% ε, του χρόνου σας. Ξεπεράσατε μάλλον, συγγνώμη, κατά πολύ τον χρόνο σας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση. Αυτή ο επόμενος ομιλητής. Εξ ονόματο του κ. θα έχω τρία συγκεκριμένα θέματα να θέξω και πέντε γενικά ζητήματα. Καταρχά, είναι σημαντικό να αυξηθεί ο συνολικό ε, προπολογισμό του Horizon Europe. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ε, έρευνα για το διάστημα, θα πρέπει να υποστηριχθεί στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Και τρίτο συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να συμμετέχει. Μπορεί ε, να συμμετέχει η Ελβετία και το Ισραήλ, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και το Εμένο Βασίλειο. Πέντε γενικά θέματα τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μόνο ένα μικρό τμήμα του συνολικού προγράμματο έρευνα και ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε λοιπόν να πιέζουμε τα κράτη-μέλη που δεν ε, δαπανούν το 3% να το πράξουν. Και επίσης, δύο τρίτα τη έρευνα και ανάπτυξη δεν είναι από τι δημόσιε δαπάνε, αλλά από ιδιωτικέ δαπάνε, από τι εταιρείε. Θα πρέπει να δαπανούν τα χρήματα αυτά. Κατά τρίτον, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ιδεολογία με επιστημονικά τεκμήρια. Είδαμε πρόσφατα κάτι τέτοιο με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά βλέπουμε ότι ισχύει αυτό και στο κοινοβούλιο. Έχουμε πολλέ παραβιάσει των επιστημονικών τεκμηρίων προκειμένου να υποστρέψουμε αναπτυχθεί η πολιτική ατζέντα του καθενό Κατά τέταρτον, ο προηγούμενο ομιλητή, το είπε η προηγούμενη ομιλητρία. Δεν θα πρέπει να μειώσουμε τι επενδύσει στα κοινωνικά θέματα. Αυτό επαναλαμβάνεται διαρκώ, Δεν μιλάμε μόνο για την τεχνολογία. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Και τέλο, υπάρχει το R, υπάρχει και το D η έρευνα και η ανάπτυξη. Θα πρέπει να επιτρεθούμε στην έρευνα. Γιατί τίθεται το θέμα του συστήματος ε, ελεύθερης αγοράς. Αυτό δεν προωθεί τις μακροπρόθεσμες ε, επενδύσεις από τις εταιρείε. Αυτό είναι πρωταρχικά ρόλος του κράτους. Θα πρέπει να υπάρχει επικέντρωση λοιπόν στη βασική έρευνα και να απόσχουν από θέματα ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Η κυρία από την Άλτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις επιτρέψτε μου. Ε, για την ομάδα μου, τους φιλελεύθερους, η αριστεία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζητμίο. Η αριστεία, λοιπόν, θα φροντίσει προκειμένου να προωθηθεί η επιστήμη μας και να είμαστε ανταγωνιστικοί στον κόσμο. Ε, πέραν τούτου, όπω είπαν οι συνάδελφοι, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πληρούν τι προποθέσει και τι συμφωνίε οι οποίε έχουν γίνει Έχουμε πει λοιπόν 30%, 30 έρευνα και ανάπτυξη. Σχεδόν κανένα κράτος μέλος δεν τηρεί αυτό το 3% και θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό στους κόλπους του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα ευθυντικά ταμεία. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό τα ευθυντικά ταμεία να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του Horizon Europe σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί και που ορίζονται από τα κρατημέλη. Και τα προγράμματα με σφραγίδα αριστείας να μπορούν να υπολογίζουν στη χρηματοδότηση αυτή. Και είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά την ε, κρατική επιδότηση. Το, η έκκληση να αυξηθεί το ποσό σε 120 εκατομμύρια είναι πολύ σωστή και είναι πολύ σημαντικό να λυθούν οι αποφάσει αυτέ για το μέλλον, για την βασική έρευνα, τη θεμελιώδη έρευνα. Το τονίζω αυτόν τον όρο, γιατί μπορεί να έχει μεγάλη πιθανότητα αποτυχία, αλλά ουσιαστικά δημιουργεί τι βάσει για το μέλλον. Μετά το Horizon Europe, το, το μέλλον το οποίο θα πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε να οικοδομούμε με την θεμελιώδη έρευνα και σε συνεργασία με την ε, βιομηχανία η συνεργασία με τη βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου όχι μόνο να έχουμε συνεργασία, αλλά και οικονομική συνεισφορά για την κοινοτομία και την έρευνα που σημειώνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η συνέργεια, γιατί όντω αυτό θα μας δώσει ανταγωνιστική χρειά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντελίντε, το IPCC προσφάτως δημοσίευσε μία έκθεση όσον αφορά το κατεπήγον της κλιματική αλλαγή. Ο δημοσιογράφος του BBC είπε τα εξή ε, από τους επιστήμονες προς πολιτικού. Τρει λέξει. Ε, ε, αντιδράστε αμέσως ανόητοι και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με τον ορίζοντα Ευρώπη, να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό τη έρευνα. Ε, και της καινοτομίας για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις αλλαγές ε, που ε, είναι αναπόφευκτες στον ορίζοντα μέχρι το 2030. Δώσαμε έναν προϋπολογισμό δώσαμε έναν προπολογισμό τον οποίο είχαμε συσχετίσει με έναν στόχο, τον οποίο χάσαμε, λέει το ελεγκτικό συνέδριο, κατά 5%. Ε, τελικά δηλαδή η συνεισφορά μας στην άμβληση της κλιματικής αλλαγής δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Πρέπει να αυξήσουμε τον προπολογισμό ε, για ε, την κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε προπολογισμό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουμε τους στόχους μας και την απαραίτητη, τους απαραίτητους κανονισμούς, την απαραίτητη ρύθμιση, ώστε να μας επιτρέψει να ε, προβούμε στα απαραίτητα μέτρα, να επιτύχουμε το στόχο μας ε, και να έχουμε και τον απαραίτητο ε, προπολογισμό. Εσάς, ποια είναι η εκτίμησή σας αυτής της έκθεσης του IPCC, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να απελευθερώσει όλο αυτό το δυναμικό και να εκπληρώσει τους, τους, τις υποχρεώσεις της από τη Συμφωνία των Παρισίων. Ε, η Γκουε τώρα. κανένα από τους ε, αξιότιμους συναδέλφου δεν είναι εδώ. Οπότε εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Στον ορίζοντα Ευρώπη πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τις μεταφορές και ε, το, τα διαστημικά προγράμματα ε, που είναι κάτι το οποίο μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει, δηλαδή τα διαστημικά προγράμματα μπορούν να μας βοηθήσουν και στις μεταφορές. Είναι πολύ συνδεδεμένα αυτά. Επίσης, τα μικρο σωματίδια που είναι επίση πάρα πολύ σημαντικά όχι μόνο στους τομεί της βιομηχανία, αλλά και για την υγεία μας. Τρίτος τομέας, η βιολογία. Νομίζω ότι δεν ε, χρειάζεται ιδιαίτερη αξιολόγηση αυτό, το γνωρίζετε και μετά υπάρχουν και τα κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα. Έχουμε πάρα πολλές ε, νέες ε, προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε ε, και μάλιστα οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ ταχείες, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να αφιερώσουμε ένα τμήμα των προσπαθειών μας στο σχετικό κομμάτι της έρευνας και βασικής έρευνας όσον αφορά τώρα τη σωστή ισορροπία μεταξύ της βασικής και της περαιτέρω έρευνας, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ισορροπία. από 100 σε 120 δισεκατομμύρια ευρώ να περάσουμε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το ποσό είναι το κατάλληλο ε, για να επιτύχουμε τους στόχους μας με την έρευνα όπως είπε και η συνάδελφος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας συνδυασμός της βασικής έρευνας και της περαιτέρω έρευνας, αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας με ε, τη βιομηχανία. Ε, γιατί πρέπει να υπάρξει αυτή η σύνδεση. Αυτά είναι τα δικά μου σχόλια και δεν εξάντλησα τα δύο μου λεπτά. Τώρα... Η κυρία Νταμάτο δεν είναι εδώ. Κυρία Κόπελ. Έφυγε. Η κυρία Κατάινεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία λεπτά νομίζω ότι έχω, γιατί είμαι εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Αγαπητοί εισηγητέ και συνάδελφοι, ένα τόσο ισχυρό πρόγραμμα, ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα πλαίσιο χρειάζεται για να υποστηρίξουμε την αριστεία ε, στην έρευνα και την καινοτομία. Αυτό ο μεγαλύτερο προπολογισμό είναι βεβαίω ε, πολύ ευπρόσδεκτος βελτιώνει πολύ επιτυχώς το πρόγραμμά μας ε, Horizon Ευρώπη. Εγώ ε, η συγγήτρια της Επιτροπής Γεωργίας θα ήθελα να αναφερθώ ε, στην, πέμπτη ομάδα που έχει να κάνει με τη φύση και τους φυσικούς πόρους τα 10 δισεκατομμύρια που χρειάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Η ασφάλεια ε, των τροφίμων ε, δεν είναι κάτι το αυτονόητο γιατί υπάρχει κλιματική αλλαγή που αποτελεί μία πρόκληση ε, και οι επενδύσεις δεν είναι επαρκείς πάνω από 800 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο υποφέρουν από υποσυτισμό. Επίσης, ε, από 12 φυτά προέρχεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ε, τμήμα των, ε, της διατροφής των ανθρώπων παγκοσμίω. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Φυσικά η αύξηση του προπολογισμού είναι ένας καλός τρόπος όταν προσπαθούμε να βρούμε βιώσιμους τρόπους καλύτερης χρήσης του περιβάλλοντος. Θα ήταν χρήσιμο όμως να υπάρχει και εφαρμοσμένη επιστήμη που θα χρησιμοποιείται. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Νίκα Είπε δηλαδή ότι σε επίπεδο εφαρμογής πρέπει να υπάρχει έρευνα. Αυτό σημαίνει δηλαδή και επιχειρηματικότητα, να συμπεριληφθούν και οι γεωργοί, να υπάρχει δηλαδή και μια ε, έρευνα που θα γίνεται επιτόπου. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο προσέγγισης ε, της ε, κυκλικής οικονομίας να λάβουμε υπόψη, ε, για παράδειγμα, ε, την γεωργία, τη δασοκομεία, για να αντικαταστήσουμε τα πλαστικά, για παράδειγμα. Δεν μιλάω μόνο για τους ωκεανούς και τις θάλασσες. Πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και τις εσωτερικές πλωτές οδούς μας ε, και τις λίμνες μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με άλλα προγράμματα. Αυτό Ήδη έχει συζητηθεί η ομάδα 5 πρέπει να αναδιατυπωθεί προκειμένου να ληφθεί η υπόψη, να, να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της κοινή γεωργικής πολιτικής που αλλάζουν συνεχώς και που τονίζουν τη σημασία της έρευνας και ελπίζω ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας θα ληφθεί υπόψη, ειδικότερα όσον αφορά την ομάδα αυτή 5 και ότι το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την διάθεση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ε, ώστε να διατηρηθεί αυτός ο προπολογισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 10% ε, μόνο, κατά 10% ε, ξεπεράσατε το χρόνο σας, παρά το γεγονός ότι είστε εισηγήτρια. Σας άφησα πάντως να μιλήσετε λίγο παραπάνω. Ο κύριος Φανίστελ Ρόι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Όχι για να προβώ σε αυτόν τον κανιβαλισμό που αναφέρατε, αλλά για να συνεισφέρω στη συζήτηση. Τι συνέβη στην περιφερειακή πολιτική. Την αλλάξαμε. Υπάρχει αιρεσιμότητα Επτά χρόνια πρώτη, το, το πρώτο και μεγαλύτερο τμήμα των 48 δισεκατομμυρίων αφορούσε την έρευνα και την καινοτομία. Ήταν μια σιωπηρή επανάσταση στον τομέα Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε για παράδειγμα ένα πολύ μεγάλο Airbus, αλλά πρέπει να έχουμε και έναν αεροδιάδρομο για να προσγειωθεί. Γιατί είναι ζήτημα κυριότητας. Υπάρχει συχνά μια εδαφική πτυχή, μια εδαφική διάσταση, τον τρόπο με τον οποίο ας πούμε ε, εκπαιδεύουμε τους μηχανολόγους μας ε, ε, και Γι' αυτό ακριβώς συχνά είναι ευφυή η περιφερειακή μα πολιτική. Δεν μπορεί κανείς να είναι καλό σε όλα. Είναι σημαντικό λοιπόν τα κράτη-μέλη από κοινού με τους εταίρους τους να κάνουν μία επιλογή από όλες τις εναλλακτικέ επιλογές που έχουν ε, και γι' αυτό σε αυτό το σημείο μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς. Εγώ είμαι εισηγητή και λέω ναι στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να χρησιμοποιήσει αυτό το 5% να φτάσει στον ορίζοντα Ευρώπη ή αντιστρόφως για να είναι καλύτερα τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας ε, στις περιφέρειες, στις πόλεις, στην εδαφική διάσταση εν πάση περιπτώσει όχι να έρθουν τα χρήματα πρώτα στι Βρυξέλλε, απευθείας ε, να διατεθούν τα χρήματα στι περιφερειακέ δραστηριότητες, ε, εκεί όπου γίνεται η καινοτομία. Και αυτό είναι το τρίτο τμήμα του προγράμματός σα. Ε, είναι το να γίνονται τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Ο κύριος Κένκελ είπε για παράδειγμα ότι δεν είναι, ότι, είπατε ότι δεν, ε, δεν υπάρχει επιλογή. Πρέπει όμως να υπάρχει επιλογή και να λέμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα την καινοτομία. Η δυσκολία είναι, οι νέοι είναι ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. 50% είναι στην Πολωνία οι νέοι του πληθυσμού. Αυτά είναι τα κύρια κέντρα της αριστείας όπου ο νικητής κερδίζει τα πάντα Έχουμε πάρα πολύ δυναμικό και θέλουμε το 1 πέμπτο του προπολογισμού μας να συνεχίσει να αφιερώνεται ε, με τρόπο από πάνω προς τα κάτω, να είναι αντικείμενο πούμε, κεντρικής διαχείρισης, με όποιο τρόπο θέλετε. Εγώ θα υποβάλω την έκθεσή μου εγκαίρως, ώστε να ε, το λάβετε υπόψη. Εμείς υποστηρίζουμε τη σφραγίδα της αριστείας, ε, ε, είμαστε υπέρ της χρήσης της για να μπορέσουμε να αυξήσουμε και την απασχόληση. 10% ξεπεράσατε κι εσείς το χρόνο σας, όπως και η προηγούμενη συγκήτρια. Άλλοι συνάδελφοι τώρα θα πάρουν το λόγο. Η κυρία Κουμπούλα Νάτρη. Δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σα. σα ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και προσπαθήσω να σεβαστώ το όριο. Νομίζω ότι η αριστεία είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους γιατί πρέπει να επιλύσουμε δύσκολα προβλήματα και δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε παρά μόνο αν είμαστε οι καλύτεροι. Θα χρειαστούμε λοιπόν αυτή την ε, κορυφαία έρευνα στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν τα εργαλεία αλληλεγγύη τα οποία και χρειαζόμαστε για να δούμε ότι για να υπάρξει απάντηση στις κορυφαίες προκλήσεις χρειαζόμαστε και κορυφαίους επιστήμονες. Τονίζουμε εκ νέου ως κοινοβούλιο Θυμάμαι ότι στη Φλανδία, στο Κοινοβούλιο, λέγαμε ότι είναι αδύνατον να περικόπτουν τους προπολογισμού τους ε, οι κυβερνήσεις και οι χώρες και να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξάνει τον προπολογισμό της. Αν θέλουμε λοιπόν πιο πολύ έρευνα, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιο πολύ. Επίσης, ε, το μήνυμα του κυρίου Νίκα είναι ότι θα πρέπει να μιλήσουμε στον κόσμο. Η πρόκληση του Ελσίνκη, όπως ονομαζόταν από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη για παροχή δωρεάν συμβουλών. Έχουμε για καταρχάς ε, τους στόχους για τις εκπομπές, έχουμε τις ε, ομάδες διαφορετικών επιστήμονων που συνομίλησαν με πολιτικούς, με δωρητές και συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε ως ε, πολιτικοί, ως απλοί πολίτες τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Θα ήθελα λοιπόν να συμπεριλαμβάνεται η διάσταση αυτή. όχι μόνο λοιπόν να μιλάμε για την επιστήμη, αλλά να μιλάμε και με τους επιστήμονες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους ζήτησαν το λόγο και να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της ε, ακρόασής μας. Και μετά θα έχουμε γύρω ερωτοπαντήσεων. Το λόγο έχει η κυρία, ο κύριος Ντομινίκ Γκέλεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όμως θα μιλήσω στα αγγλικά, γιατί τα γνωρίζω εξαιρετικά. Έχουμε κάποια θέματα στην παρουσίασή μου. Κάποια ζητήματα από τα οποία ακούσαμε και στη συζήτηση. Θα ακούσουμε διάφορα νέα στοιχεία. Θα συζητήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα το Horizon Europe. Σχέσεις με την Ιαπωνία, Κορέα, ΗΠΑ. Και έχουμε και κάποια διδάγματα να αντλήσουμε από τη γενικότερη αυτή βάση γνώσης που έχουμε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες αρχές και το κατά πόσον μπορούν να επηρεάσουν την κατεύθυνση της ε, καινοτομίας. Ακριβώς αυτό αφορά το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Κατά δεύτερον, η θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Και τρίτον, ε, διακυβέρνηση και προσανατολισμός του Horizon Europe. Λυπάμαι είναι μεγάλη η οθόνη, αλλά δεν φαίνεται καλά η διαφάνειά μου. Είναι μεγάλη η αθούσα. Δαπάνες ε, δημόσιες για την έρευνα και την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις ε, από τα τέλη του 2008 από την ε, οικονομική κρίση τελμάτως ουσιαστικά και μείωση των επενδύσεων, των δημόσιων επενδύσεων, ενώ οι δαπάνες από τις εταιρείε αυξάνονταν. Αυτά στον ΟΑΣΕ. Κοιτώντα τώρα πιο συγκεκριμένα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς είναι, ίδια είναι η τάση τελμάτωση των ε, κρατικών επενδύσεων και αύξηση των επενδύσεων από πλευρά των επιχειρήσεων. Σε επίπεδο χωρών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιλέξαμε τις χώρες οι οποίες ταπανούν πιο πολύ στην έρευνα και ανάπτυξη. Όλες οι χώρες στο γράφημα, εκτός από την κάτω-κάτω που είναι η Σουηδία, σημείωσαν τελμάτωση ή και σημαντική μείωση σε ό,τι αφορά τη θέση του στην έρευνα και ανάπτυξη. Συνολικά λοιπόν διαπιστώνουμε μείωση 3 έως 4% σε ό,τι αφορά τις κρατικές ε, δαπάνες ε, και στην έρευνα και την ανάπτυξη. Φυσικά γνωρίζουμε ότι τα χρήματα δεν επιλύουν όλα τα προβλήματα, αλλά προφανώς έχουν αντίκτυπο. Η μείωση λοιπόν της χρηματοδότησης ε, σημαίνει μείωση της επιρροής. Και ακόμα χειρότερα σε κάποιες περιπτώσεις, κοιτώντα κάποιες ε, συνοριακές τεχνολογίες και η κυρία Καλίτσκα αναφέρθηκε στην ε, τεχνητή νοημοσύνη, εδώ οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες δαπάνες απουσιάζουν. Ε, Επί 40-50 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη ήταν μόνο στα χέρια της κυβέρνησης ε, των πανεπιστημίων. Τώρα όμως έχει περάσει στα χέρια αποκλειστικά των επιχειρήσεων. 30-40 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανούνται για την ε, τεχνητή νοημοσύνη και η μηδενική είναι η συμμετοχή ουσιαστικά των ε, κυβερνήσεων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ουσιαστικά την κατεύθυνση καθορίζουν οι επιχειρήσεις. Αυτό προφανώς και οδηγεί σε βασικές ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την ικανότητα, τη δυνατότητα των κρατών να προσανατολίζουν, να καθοδηγούν τις εξέλιξεις. Μπορεί να ισχυριστείτε ότι υπάρχουν φορολογικά πλέον Είναι σημαντικό το σκέλος αυτό. Δεν το έχω συμπεριλάβει στην ε, παρουσίασή μου, αλλά τα φορολογικά κίνητρα ουσιαστικά δεν δίνουν κατεύθυνση στην έρευνα και την ανάπτυξη. Δεν επηρεάζει τις ε, επιλογές βάση που λαμβάνουν χώρα βάσει της αγοράς. Άρα χάνει την επιρροή της ε, η κυβέρνηση. Αυτό να το έχουμε υπόψη ότι είναι μειούμενη η επιρροή που ασκούν οι κυβερνήσεις. Στη συνέχεια, το μειούμενο ε, μερίδιο της ε, Ευρώπης στο παγκόσμιο προσκήνιο. Βλέπετε στο γράφημα και άλλες ε, περιοχές της ΙΠΑ, την Ιαπωνία και το καθεξής. Αν συγκρίνουμε τους οικονομικούς όρους αν συγκρίνουμε λοιπόν τα προγράμματα πλαίσιο με τα μεγάλα προγράμματα στον κόσμο, στον ΙΠΑ το NIH είναι 32 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα και το NSF, το οποίο εκτελεί μόνο θεμελιώδη έρευνα στη ΣΥΠΑ. 6 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό τι σημαίνει ότι το Horizon Europe είναι σημαντικό. Δεν είναι μικρό ποσό, αλλά δεν είναι και κάτι ε, εξαιρετικό. Να μην ε, υπερεκτιμούμε το τι μπορούμε να πετύχουμε με τα χρήματα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας εξετάσουμε τώρα και κάποιους άλλους όρους για το Horizon Europe προκειμένου να δούμε τι μπορεί να πετύχει πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο. Καταρχάς, να μην έχουμε υπόψη μας μόνο την έρευνα, αλλά και τους συμπληρωματικού όρους, προκειμένου να είναι επιτυχής η δαπάνη στην έρευνα. Στην Ευρώπη έχουμε ένα πρόγραμμα πλαίσιο για τους Ευρωπαίους. Και κατά τα άλλα έχουμε 28 ουσιαστικά χώρες, 28 αγορές για τα προϊόντα. Είναι τεράστιο το κόστος προφανώς για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις νεοφύης. Άρα, ο, σε ό,τι αφορά τον πραγματισμό ενεργειών και δράσεων, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κεφαλαγορά δεν υπάρχει ουσιαστικά ιδιαίτερα και για τα venture capital και εν ώψη του Brexit, καταλαβαίνετε, μιας και το Λονδίνο, το City, είναι το κέντρο του venture capital στην Ευρώπη. Το μέλλον της ε, τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αγορά για τα δεδομένα. Γίνονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή και στο Τάλιν πέρσι έγινε μια σημαντική σχετική προσπάθεια, αλλά κοιτώντα το δρόμο που έχει διανύσει ακόμα η Ευρώπη, τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι μακρύς ο δρόμος. Μπορούμε να δαπανίσουμε λοιπόν πολλά χρήματα, σημαντικά ποσά. Αλλά αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι όροι και οι συνθήκες για να ανθίξει ο κλάδος ε, της έρευνας, δεν θα καταφέρουμε και πολλά. Α, αναφέρθηκε το πρόβλημα των ε, στόχων ε, και της πολυσυμφετότητας των στόχων σε ό,τι αφορά τους στόχους, τους βιώσιμους στόχους, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την αριστεία, σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί ενδεχομένω να μην ε, συνάδουν απαραίτητα πάντα όλοι οι όροι αυτοί, αλλά υπάρχει πάντα, για παράδειγμα, αυτή η διαφορά μεταξύ αριστείας και της ε, συμπερίληψης. Είναι πολύ λοιπόν και διαφορετική η στόχη, είναι πολύ και διαφορετική και οι εμπλεκόμενοι φορές. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την επέκταση του αντίκτυπου ενός προγράμματος. Χρειάζεται να υπάρχει μόχλευση των εθνικών δαπανών. Όπως σας είπα, το πρόγραμμα πλαίσιο είναι το 10% των δημοσίων δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. 90% προέρχεται από τις εθνικές κυβερνήσεις, άρα βάσει του προγράμματος πλαίσιο δεν θα προχωρούσαμε ιδιαίτερα. Και τέλος υπάρχει αυτή η συζήτηση μία μόνιμη συζήτηση για τη διαφορά της ε, θεμελιώδους ε, και της εφαρμοσμένης έρευνας. Να αναφέρω. Κάτι το οποίο δημοσιεύτηκε και σε ένα βιβλίο πριν από 20 χρόνια. Δεν υπάρχει ουσιαστικά διαφορά μεταξύ των δύο τύπων έρευνας. Χρειαζόμαστε και τα δύο. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποια επιτυχία, αλλά η βασική αυτή έρευνα μπορεί να ενταχθεί και στις αποστολές. Αν θέλουμε μακροπρόθεσμο αντικτύπο, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνο βραχυπρόθεσμοι στόχος. Άρα η βασική έρευνα θα πρέπει να ενταχθεί στα προγράμματα αυτά. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Αν θέλουμε να αυξήσουμε λοιπόν τον αντίκτυπο ενό προγράμματο το οποίο δεν είναι πολύ εκτενέ, θα πρέπει να λεφτούν συμπληρωματικά μέτρα. Θα πρέπει να υπάρχουν εταιρικέ σχέσει και συνοχή με τα εθνικά προγράμματα και με τα εταιρικά προγράμματα και θα πρέπει να ενταχθεί η βασική έρευνα στην καρδιά, στον πυρήνα των προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κελέκα. Τελευταίος ε, στον κατάλογό μου είναι ο προκαθηγητής Γιάννος Βιλέξκη. Thank you, Mr. Chair. Ε, members of the e Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ήτρε, πρώτα απ' όλα ε, να απαντήσω σε μια ερώτηση που ήταν στη διάρκεια της συζητήσεως. Πού είναι ο Ευρωπαίος πολίτης στον κύκλο της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων κλπ. Κάπου εκεί. Πολλά στοιχεία που αναφέρθηκαν είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πούμε η έκθεση IPC, η οποία παρουσιάζει τεκμήρια επιστημονικά ότι οι επιστήμοι και οι επιστήμονες καλά έκαναν τη δουλειά τους και ίσως τώρα πρέπει και οι πολιτικοί να αναλάβουν δράση ε, επομένως, ε, η ερώτηση θα έπρεπε να διατυπωθεί διαφορετικά. Πού είναι ε, οι policy makers, πού είναι αυτοί οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν την πολιτική βάση των οδηγιών των επιχειρηματιών. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω ως επιστήμον και λέω ότι πρώτα απ' όλα το πιο σημαντικό είναι να βρούμε ποιες είναι οι αποστολές τις οποίες θα πρέπει να καλύψουμε και με ποιο τρόπο θα καλύψουμε τις αποστολές. Στη διαδικασία αυτή το σημαντικό είναι να συμπεριληφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εξ αρχής να γίνουν συνεργασίες. Επομένως θα πρέπει και η κοινωνία των πολιτών και τα κράτη-μέλη και η κοινωνία των ε, ερευνητών να συμπεριληφθούν και όσο γίνεται πιο ε, σαφώς να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα ε, συνεργαστούν και ε, ακολουθώντας και κάποια παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν ήδη μπορούν να υπάρχουν συγκεκριμένες συνεργασίες συμπεριληπτικές οι οποίες ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, αλλά ε, η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων θα πρέπει να ξεκινήσει από την εδρεωμένη ε, έρευνα σε χαμηλότερο επίπεδο και για συγκεκριμένα θέματα. Το σημαντικό επίσης είναι και η προτεραιότητα είναι να υπάρχει προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, άρα αντιμετώπιση συνολικών ζητημάτων με συμπεριληπτικό τρόπο. Όσον αφορά τα εργαλεία, τα grants ε, θα πρέπει να παραμείνουν ε, το κεντρικό εργαλείο για την ε, χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας και στους τρεις πυλώνες και την Open Science και τις συνολικές προκλήσεις αλλά και την ανοιχτή καινοτομία. Θα πρέπει οπωσδήποτε και στα τρία, στους τρεις πυλώνες να δίνονται αυτές οι υποτροφίες και όχι μονάχα στα πλαίσια του ε, ERC. Όπως και στον, στο δεύτερο πυλώνα ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθηθούν συμπεριληπτικά προγράμματα, ε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και να υποστηριχθούν βεβαίως όλα τα επίπεδα από το επίπεδο 1 μέχρι το επίπεδο 8 και αυτό στα πλαίσια του πυλώνα 2 και ε, επίσης εξαιρετικά σημαντικό είναι να απλουστευθούν οι διαδικασίες όταν κάποιος ζητάει ε, μια υποτροφία, ένα grant. Θα πρέπει λοιπόν αυτού του είδους η έρευνα να προχωρήσει γρήγορα μέσα από γρήγορη διεκπαιρέωση ε, και του αιτήματο για grant. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα ήθελα ε, να ε, αναφέρω γιατί σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ε, κλείσει αυτή η ψαλίδα της έρευνας και ε, ε, καινοτομία στην Ευρώπη ε, είναι μέσω της αντίληψης ότι υπάρχει ήδη η αριστεία σε πολλές χώρες και στις λεγόμενες widening countries υπάρχει ήδη αριστεία. Υπάρχουν και δίκτυα αριστείας τα οποία φαίνεται να μην θέλουν να διευρυνθούν. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι σημαντικό να διευρυνθούν τα υφιστάμενα δίκτυα ε, αριστείας γιατί δεν πρέπει να αποκλείεται κανένας, δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί όσον αφορά την ε, αριστεία. Επομένως ε, και οι δράσεις οι οποίες έχουν αναλυφθεί στα πλαίσια της προσπάθειας διεύρυνσης είναι καλές, αλλά βεβαίως θα πρέπει να ακολουθηθεί και από διεύρυνση και το, του προϋπολογισμού. Ε, ε το σημαντικό φυσικά, το ακόμα σημαντικότερο είναι το ζήτημα αυτό να θεωρηθεί ε, οριζόντιο ζήτημα στα πλαίσια του προγράμματος, αλλά βεβαίως να μην να μην ε, αποκλείονται ε, οποιασδήποτε χώρες από τη διαδικασία αυτή. Βεβαίως η αρχή της αριστείας θα πρέπει να γίνεται σεβαστή σε κάθε περίπτωση και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να ε, εισαχθούν συγκεκριμένοι στόχοι ας πούμε οι οποίοι θα βασίζονται και σε πολιτική συμφωνία ε, π.χ. συγκεκριμένοι στόχοι για την αύξηση συμμετοχής από το 4% στο 10%. Αυτό μπορεί να αποτελεί έναν σαφή στόχο σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ε, και μπορεί να αποτελέσει ένα απολύτημα, απο, απόλυτα συγγνώμη, μετρήσιμο δίκτυο συμφωνώ με ε, ε, αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, ε, δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει κινητροδότηση στους, ε, στις συμπράξεις και τους ομίλους έτσι ώστε να διευρύνουν κατά κάποιο τρόπο το είδος των συμμετοχόντων. Ωστόσο πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε αξιολόγηση που θα βασίζεται στην αριστεία αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι τα κριτήρια επιλογής μπορούν να τροποποιηθούν ε, και οι οι ε, προτιμήσεις ε, καθώς επίσης και η ιεράρχηση να ε, είναι πλέον πιο διαφορετικές. Θα πρέπει να εστιάσουμε πάντως στην μέχρι τώρα εμπειρία μας γιατί ορισμένοι μηχανισμοί έχουν λειτουργήσει. Μην το ξεχνάμε αυτό πάντα όσον αφορά την ε, μοιρασμένη αριστεία πιστεύουμε ότι οι συνέργειες θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω ε, και να ε, εκμεταλλευτούμε κυρίως αυτές οι οποίες έχουν σχέση με τα διορθωτικά ταμεία τα οποία ακριβώς αφορούν τις περιφέρειες. Ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό που υπόθηκε προηγουμένως εδώ, κανιβαλισμός. Δεν θα πρέπει να κανιβαλιστούν δηλαδή οι ε, καλοί μηχανισμοί και αυτοί που λειτουργούν σωστά. Κοιτάξτε, μην λησμονούμε ότι τα διευθυντικά ταμεία αφορούν τις περιφέρειες, τα προγράμματα απευθύνονται στα κράτη. Επομένως θα πρέπει απλώς όχι να μπερδέψουμε τα πράγματα, γιατί με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ε, και κακή κινητροδότηση βάσει του εσωτερικού ανταγωνισμού, αλλά θα πρέπει ενήθως να δημιουργήσουμε ε, καλές συνέργειες. Οπωσδήποτε ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει επικάλυψη των μηχανισμών και θα πρέπει ε, η διεύρυνση να βασίζεται στους ε, δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα Horizon 2020. Όπως ε, είπα και προηγουμένως, ε, θα πρέπει η χρηματοδότηση ε, των προγραμμάτων που έχουν τη σφραγίδα της αριστείας να βασίζεται στους κανόνες του Horizon Europe, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων για κρατικές επιδοτήσεις. Εγώ τώρα ήθελα να θίξω κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν ήδη χρηματοδότηση των ερευνητών. Βεβαίως υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην αίσθηση του ε, αντικτύπου που δεν βασίζεται ε, και δεν αντιπροσωπεύει ακριβώς ε, το είδος της αριστείας αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας νέος μηχανισμός έτσι ώστε οι μηχανισμοί των widening states να μπορέσουν να ανταγωνιστούν σε ίσο επίπεδο και επομένως να υπάρχει καλή συνέργεια ανάμεσα στα εφιστάμενα δίκτυα και τα δίκτυα που προσδοκούν να βελτιωθούν. Εξαιρετικά, λέει ο πρόεδρος. Δεν ξεπεράσετε καθόλου το χρόνο σας. Μπράβο σας και έβγε σας. Λοιπόν, Ο κύριος Νίκα πρώτος ε, να μας πει τι παρατηρήσεις του για το δεύτερο τμήμα των ε, παρουσιάσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους εισηγητέ και όλους τους ομιλητές. Τονίσατε τα κριτήρια της αριστείας, ότι δεν είναι αριστεία έναντι της ε, επέκτασης, της διεύρυνσης ε, του προγράμματος. Θα ήθελα να πω κάτι για την προηγούμενη μου παρέμβαση. Κάποιος με ρώτησε τι γίνεται με το γεγονός ότι δεν έχουμε χρήματα να δώσουμε σε όλο τον κόσμο. Να διευκρινίσω. Εγώ αυτό που είπα κυρίως ε, ήταν ε, να αναφερθώ σε κάποιες ιδέες που υπάρχουν ότι πρέπει να βοηθήσουμε την, ε, την Κίνα. 18% τον, ε, της χρηματοδότησης πηγαίνει σε Κινέζους ε, γιατί δουλεύουν στο ΕΡΑ ε, για, κάποια, για κάποιο πρόγραμμα. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται μετά αν φύγουν αμέσω μετά, εμεί με τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της κινεζική οικονομίας και όλοι σα μιλήσατε για την αντιπαραβολή της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πολύ σαφείς κανόνε αν είναι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πώς θα τα δώσουμε αυτά τα χρήματα και να υπάρχουν κρατήρια. Αν κάποιος υπήκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα, κάνει ένα διδακτορικό για παράδειγμα ε, σε κάποιο πανεπιστήμιο, όποιο πανεπιστήμιο τον φιλοξενεί πρέπει νομίζω να παραμείνει στον φορέα αυτό και μερικά χρόνια αφού του τελειώσει ε, η υποτροφία, η χρηματοδότηση, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία συνεισφορά στον απότερο στόχο μας που είναι να έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο παίκτη και να έχει μια καλύτερη θέση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Όσον αφορά αυτό το widening, ε, λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν αξιολογητές ε, και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων από όλες τις χώρες και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εγώ έρχομαι από μια χώρα που είναι καθαρός εισφορέας ε, για τον ορίζοντα 2020 ε, μας είπαν οι δωρητές, ε, δικά μας είναι τα χρήματα, πρέπει να έχετε τους ανθρώπους μας στο διοικητικό συμβούλιο. Ε, δεν πρόκειται να πάρετε τα δικά μας τα χρήματα και να τα κάνετε ό,τι θέλετε, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Το ίδιο πράγμα λέω κι εγώ. Αν θέλουμε να είμαστε μία από τις χώρες δωρητές, πρέπει να έχουμε κι εμείς την άποψή μας που θα μετράει. Θα πρέπει ο βασικός επιστήμονας να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο για να κάνει την αξιολόγηση. Διαφορετικά υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό σε σχέση με το τι θα γίνει μετά. Θα σταματήσω εδώ. Δεν θέλω να δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ώστε για να μπορέσουμε να, μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα, όλες τις αδυναμίες πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια και όλοι πρέπει να δουλεύουν επί τη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων ε, το EIC για παράδειγμα θα θέλα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία ακόμη φορά να σκεφτεί ε, έναν τρόπο, δεν έχω εγώ την νομική ε, τεχνογνωσία τι θα μπορούσε να είναι το, ο μεγαλύτερος φόρτος για το ΕΣΥ. 20% ποσοστό επιτυχίας πρέπει να έχει. Τουλάχιστον αν δεν υπάρχει αυτό γραμμένο κάπου με νομικούς όρους θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί το ελεγκτικό συνέδριο θα ζητήσει 100% ποσοστό επιτυχίας ε, γιατί πρόκειται για χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω αυτό για να κάνω μια διευκρίνηση ε, σε σχέση με το που βρισκόμαστε. Έχουμε και πολλές ε, άλλες ε, συνεδριάσεις οδών. Κάναμε μία ήδη, θα κάνουμε και άλλες τρεις. Έχουμε λοιπόν χρόνο να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση η οποία θα είναι ε, εποφελής και για σας τους ερευνητές και για μας ε, ως πολιτικούς. Αν εσείς είστε ευχαριστημένοι, είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι. Α, και κάτι άλλο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μη το βάλετε στον ίδιο κορβανά με, το, με τις συνδεδεμένες χώρες. Είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκθεση αυτή. Όταν λέμε λοιπόν ότι το ERA είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, είναι όντως συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου ε, μαζί με την Ισλανδία και την Νορβηγία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε ε, όχι μόνο οι επιστήμονες αλλά και όλοι οι ε, άνθρωποι που λαμβάνουν μια εκπαίδευση. Ε, εμείς για παράδειγμα στην Τσεχία ε, εκπαιδεύουμε Αυστριακούς και Γερμανούς ε, που εποφελούνται από το διδακτορικό ιατρικής μας και το 1 τρίτο φεύγει μετά από την Τσεχία και πηγαίνει αλλού. Δεν ισχύει λοιπόν μόνο για τους επιστήμονες, ισχύει γενικώ για ανθρώπους που έχουν λάβει μια πανεπιστημιακή μόρφωση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Καπεσόν Ρουίς, που είναι η σκιώδη εισηγήτρια των Σοσιαλδημοκρατών. Έχετε το λόγο. Μου δίνετε το λόγο. Ε, λοιπόν, και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που δεν αναφερθήκε εδώ και μου φαίνεται σημαντικό το θέμα του ε, ε γένους ε, του φίλου. Ε, πραγματικά θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ε, ε, συστάσεις, μάλλον έγιναν κάποιες συστάσεις και αυξήθηκε το ποσοστό των γυναικών, κυρίως στο Advisory Committee, αλλά όχι στα διάφορα πάνελ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει συγκεκριμένη αναφορά εντός του προγράμματος και όχι μονάχα όσον αφορά την συμμετοχή, αλλά και όσον αφορά τις ίδιες τις μελέτες ε, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε ε, και για την ε, κοινωνική, το κοινωνικό αντίκτυπο των προγραμμάτων. Θα πρέπει όμως στα πλαίσια αυτά να δούμε και τον αντίκτυπο όσον αφορά το φύλλο. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό όταν μιλάμε για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τα προγράμματα αυτά στην κοινωνία. Όταν αναλύουμε τα προγράμματα θα πρέπει πρέπει οπωσδήποτε να μην αποτελέσουν διακριτική μεταχείριση του ενός ή του άλλου φίλου. Επίσης, Ε, υπάρχει ε, ε, κενό αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βρουν τους μηχανισμούς έτσι ώστε να συμπληρώσουν τον ορίζοντα Ευρώπη και όχι να υποκαταστήσουν. Ίσως θα έπρεπε να πούμε ε, ότι η επένδυση όσον αφορά την ε, απεικονιση 3 3D ε, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί ενώ δεν έχει συμπεριληφθεί. Εάν έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, ε, θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε μονάχα για το πώς θα το υλοποιήσουμε. Θα πρέπει να ψάξουμε συγκεκριμένα ε, παραδείγματα. Για να υπάρξει σωστή ε, συνέργεια θα πρέπει να ψάξουμε συγκεκριμένες ε, πρωτοβουλίες έτσι ώστε να τελειώσει το προηγούμενο πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη όμως όλα τα θετικά στοιχεία τα οποία από αυτό απορρέουν. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο. Η κυρία Βίρινγκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικέ πρατρήσει, επιτρέψτε μου. Δεν το συζητήσαμε ακόμα σήμερα, αλλά το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Ο παράγοντα του χρόνου. Θα πρέπει να φροντίσουμε να καταλήξουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβόλιο σε μια συμφωνία και θα πρέπει να ακολουθήσει και η Επιτροπή τελικά να μην υπάρχει κάποιο κενό, να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου να μην υπάρχει χρηματοδότηση επειδή δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση. Σας καλώ λοιπόν να φροντίσουμε όλοι μαζί να ολοκληρώσουμε το φάκελο αυτό προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί το έργο της επιστήμης και να μην κολλήσουμε σε κάποιο σημείο και να χρειαστεί να περιμένουμε χρηματοδότηση και να χάσουμε τη θέση μα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να συμμετέχει πιο πολύ ο πολίτης. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα σε αυτό το θέμα. Τα 751 μέλη του Κοινοβουλίου που έχουν όλοι ε, εκλεχθεί από τους πολίτες. Είμαστε εκπρόσωποι του πολίτη. Ήμουν και στο Μόσπονδο, λοιπόν, Κοινοβούλιο και το ίδιο ε, ισχύει και εδώ. Κατά τρίτον, ο η Ευρώπη 2020 έκαναν το έργο τους και μεταξύ άλλων δημιούργησαν και θέσεις απασχόλησης. Αυτές οι θέσεις απασχόλησης είναι για τον πολίτη. Ε, το 1 ευρώ που επενδύσαμε στο ορίζοντα 2020 είχε οικονομικό αντίκτυπο 11 ευρώ. Αυτό φτάνει και στον πολίτη. Και υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αντιμετωπίσαμε, όπως για παράδειγμα η υγεία, που είναι σε άμεση σύνδεση και επηρεάζουν άμεσα τον πολίτη. Πού μπορεί να γίνει περαιτέρω βελτίωση για τον πολίτη. Μεταξύ άλλων και στην επικοινωνία. Η επικοινωνία θα πρέπει να γίνει με πάρα πολύ εύκολο και απλό τρόπο, προκειμένου και ο απλός πολίτης να καταλαβαίνει για το τι μιλάμε. Ο πολίτης, ξέρετε, δεν τον νοιάζει πάρα πολύ να παράγουμε βιβλία και έντυπα. Θα πρέπει αυτά που συμβαίνουν να εξηγούνται με έναν απλό τρόπο που να γίνεται κατανοητό σε ένα λεπτό. Αυτό και τίποτε παραπάνω. Αυτό ζητάει ο πολιτή από την Επιτροπή, από το Κοινοβούλιο, αλλά και από τους επιστήμονες. Να εξηγήσουν οι επιστήμονες με απλό τρόπο τι κάνουν και σε τι αποσκοπεί η δουλειά τους. Και τότε θα καταλάβει ο πολίτης το τι συζητάμε. Αυτέ ήταν οι παρατηρήσει μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσει σας. Να δώσω το λόγο και στον εαυτό μου. Επειδή ετέθη αυτό το ζήτημα, πώς θα διατηρήσουμε το άνοιγμα της έρευνας από τη μία και από την άλλη τη σωστή επένδυση των χρημάτων μας, ώστε να υπάρχει προστιθέμενη αξία, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για τους Ευρωπαίους, όχι για τους άλλους, Η κυρία Κατάινεν. Second round, don't Όχι. Καλώς. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να θέσει ένα ερώτημα? Αν όχι, τώρα να δώσω το λόγο στους ομιλητές μας, στα μέλη του πάνελ. Θα αρχίσουμε αντίστροφα. Πρώτα ο κύριος Μπουινίτσκι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα της ε, συνέργειας και των διαρθρωτικών ταμείων και της ε, επέκτασης. Ένα από τα προβλήματα με κάποιες από τις πρωτοβουλίες ε, που εστιάζουν στην αριστεία και στην, στον μη αποκλεισμό ε, είδαν ότι η χρηματοδότηση άριστων ε, επιστημόνων ε, στις χώρες προς οποίες γινόταν η επέκταση ίσχυε μόνο για πέντε χρόνια και δεν υπήρχε μηχανισμός να παραταθεί η παραμονή αυτή ε, κάτι το οποίο ήταν ένα πρόβλημα για αυτούς τους άριστους επιστήμονες οι οποίοι ε, επιλέχθηκαν με ανοιχτούς διαγωνισμούς ε, στα πανεπιστήμια που θα έδιναν την χρηματοδότηση. Ένα από τα παραδείγματα λοιπόν της συνέργειας αυτής θα ήταν η χρήση κάποιων άλλων ταμείων όπως τα διαρθρωτικά ταμεία για τη συνέχιση των επιτυχών προγραμμάτων που έχουν αρχικά επιλεγεί ε, προς χρηματοδότηση για να μπορεί να μην υπάρχει δηλαδή ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους και να μην υπάρχει ο κίνδυνος ε, ε, να σταματήσει χρηματοδότηση ας πούμε ενός προγράμματος γιατί ξέρουμε ότι αν σταματήσει θα καλυφθεί η χρηματοδότησή του από τα διαδοτικά ταμεία για παράδειγμα. Ο κύριος Γκελέκ. Εμείς ε, στον ΩΣΑ βλέπουμε την αριστεία ευρύτερα. Ε, το καλύτερο πρόγραμμα που μπορεί να ισχύει για ε, το δικό μας στόχο πρέπει να υπάρχει μία ευρύτερη θεώρηση της έννοιας της αριστείας, να υπάρχει το άριστο ερευνητικό χαρτοφυλάκιο που δεν σημαίνει μεμονωμένα προγράμματα ερευνητικά, υποχρεωτικά. Υπάρχει ας πούμε μία τάση να χρησιμοποιείται όλη η έρευνα ε, για το ίδιο πράγμα, μία συγκέντρωση δηλαδή των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν τεθεί που, που, που, των ερευνητικών προγραμμάτων σε ένα συγκεκριμένο στόχο που έχει τεθεί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα σημαντικά τα οποία παραγνωρίζονται από την επιστημονική κοινότητα. Το θέμα της διαφοροποίησης λοιπόν, η έλλειψη διαφο, διαφοροποίησης, αξιολόγησης, γιατί πάντοτε από τους ομοτήμους γίνεται η αξιολόγηση. Υπάρχει και το θέμα του, της κατανομής ως προς το φύλλο της γεωγραφικής κατανομής, για παράδειγμα, των ε, ερευνητών. Υπάρχει λοιπόν ένα επίπεδο συλλογική χαρτοφυλακίου, για να το πω έτσι, και υπάρχουν συγκεκριμένα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αριστείας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χερλίτσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στην εξή ερώτηση όσον αφορά την αριστεία. Η αριστεία, να πω καταρχά, ότι είναι στην καρδιά των πάντων. Ισχύει και για την εφαρμοσμένη έρευνα. Ε, είναι ε, μια βασική αρχή η αριστεία, η οποία πρέπει να είναι φιλοδοξία σε ό,τι κάνουμε. Για τη συζήτηση τώρα ε, που επανέρχεται συνεχώς βασική εφηρμοσμένη έρευνα, εφαρμογή και ε, επίδειξη πρέπει να το καταλάβουμε αυτό ως τμήμα ε, της κοινή αλυσίδας αξιών. Είναι τμήμα μιας αλυσίδας αξιών κοινής. Πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί και για πολλά χρόνια συζητούσαμε το χάσμα καινοτομίας για παράδειγμα που υπάρχει στην Ευρώπη. Η μόνη λύση σε οποιοδήποτε σύστημα ε, επιτυχούς καινοτομίας ε, είναι ε, πρέπει οπωσδήποτε να ε, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών παραγόντων. Αυτό μας έχει διδάξει η πείρα μας. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να δω ότι υπάρχει κοινή έρευνα, κοινή ε, καινοτομία, ε, όλη αυτή η διάσταση να τονιστεί στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή σε όλα τα κεφάλαια αυτού. Υπάρχουν ήδη καλά παραδείγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, στα διορθωτικά ταμεία, τη γεωργία ή αλλού. Υπήρχε και αυτό το ερώτημα του προϋπολογισμού ε, κοιτάξτε, νομίζω είναι ζήτημα κρίσιμη μάζας. Πρέπει να επιτύχουμε τη συγκέντρωση των δυνάμεών μας, ε, να μπορέσουμε δηλαδή ε, ή οι διάφοροι κλάδοι από κοινού με τους ιδιωτικούς φορείς, ε, με ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρόνια λέμε ότι πρέπει όλοι αυτοί οι παράγοντες να συνεργαστούν και μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό με ρεαλιστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Η ταχύτητα και ο χρόνος είναι σημαντικά βεβαίως. Ε, ε, μου ζητήσατε να πω παραδείγματα. Νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε πολύ ακριβή ε, σε μια πολύ ακριβή εφαρμογή των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχετική πρόταση που έχει δρομολογηθεί. Η κλιματική μεταβολή επίσης αναφέρθηκε. Το τι μπορεί να γίνει είναι ένα πάρα πολύ σαφές παράδειγμα αυτό που υπάρχει πάρα πολύ έρευνα. Έχουμε πολλή έρευνα για την κλιματική μεταβολή, πρέπει όμως να την εφαρμόσουμε. Οι συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχουν στη διάθεσή του τεχνολογίες που αφορούν για παράδειγμα την ενεργειακή αποδοτικότητα, που επηρεάζουν την κλιματική ε, ε, αλλαγή εδώ. Πρέπει να υπάρξει εφαρμογή και ένα τελικό σχόλιο για την Κίνα. Νομίζω ότι εγώ το κατέστησα πολύ σαφές. Η Κίνα ε, λειτουργεί με έναν πάρα πολύ στρατηγικό και εστιασμένο τρόπο και όσο δεν έχουμε πραγματική αμοιβαιότητα, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη ε, αναπτύσσουμε την δική μας ισχύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε. Ο λόγο του κ. Σουλασλόσκη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω με δύο στοιχεία και να απαντήσω στα σχόλια του κυρίου Έλερ. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα πανεπιστήμια μίλησαν με μία φωνή και πάντα μιλούν με μία φωνή πριν από τη δημοσίευση του Horizon, ε, Horizon Europe και κάναμε, υποβάλαμε και μια κοινή δημοσίευση προς το Κοινοβούλιο. 30 πανεπιστήμια λοιπόν ε, που κατέθεσαν τις εμπειρίες τους. Μιλήσαμε με μία φωνή και μιλήσαμε χειρά προς τις κυβερνήσεις μας και θα συνεχίσουμε να τα λέμε αυτά, γιατί συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Έλερ. Είναι απαραίτητο εμείς από εκείνο το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο να συνεργαστούμε για να δώσουμε στην ε- επιστήμη στην Ευρώπη το χώρο που της αξίζει στην Ευρώπη. Δεν με έχουν ξανακατηγορήσει για κανιβαλισμό, τι να σας πω, πρώτη φορά. Αλλά να πω ότι εγώ πιστεύω το αντίθετο και το αντίθετο υποστήριξα το NSH θα πρέπει να καταστεί στρατηγικό στόχο σε όλο το πρόγραμμα. Αυτό γίνεται στην παρούσα φάση και δεν βλέπω γιατί να μην γίνει αυτό και στο Horizon Europe. Δεν κοστίζει τίποτα. Αποτυπώνω μόνο τη φιλοδοξία που έχουμε για το πρόγραμμα. Και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει α, σχετικό πρόγραμμα και προφανώ ο προπολογισμό θα θέλαμε όλοι να είναι πιο υψηλός. Εκτιμώ ιδιαίτερω τι συνεχιζόμενε προσπάθειε του Κοινοβουλίου να εξασφαλίσει μεγαλύτερο προπολογισμό για μα. Φυσικά και πάλι πρέπει να γίνουν επιλογέ. Και νομίζω ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν προσαρμογές μεταξύ των τμήματων του προϋπολογισμού, αλλά το βασικό στοιχείο για μας είναι η πραγματική ένταξη των κοινωνικών επιστήμων σε όλο το πρόγραμμα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να διαφωνούμε από αυτού. Το θέμα είναι το πώς θα το πετύχουμε. Πώς, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν το έθιξε το θέμα αυτό. Για τις αξίες. Για να απαντήσω και στο θέμα για την έκθεση SDP. Το IPCC επεσήμανε ότι οι επιστημονικές ανησυχίες για την εξέλιξη του κλίματος είναι δεδομένες. Θα πρέπει να τις ερευνήσουμε λοιπόν και θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ε, έρευνα. Μαζί με την Σουίσκο, για παράδειγμα, η οποία έχει άμα προωθήσει μια σειρά τέτοιων ε, ερευνητικών προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είναι αυτή που συντονίζει πολλά από τα ερευνητικά προγράμματα σε ό,τι αφορά την επιστήμη και επεσήμανε ότι η έκθεση IPCC επεσήμανε ότι υπάρχει όλο και πιο μεγάλο κενό μεταξύ της πολιτικής και του που βρίσκεται το IPCC. Αυτό μας επαναφέρει στο θέμα των αξιών. Ως κοινωνία λοιπόν, τι είδους εξελίξεις αντιμετωπίζουμε, ως οικονομία τι είδους εξελίξεις αντιμετωπίζουμε. Αν δεν συμμετέχουν οι πολίτες, ανησυχώ. Ανησυχώ ιδιαίτερως ότι οι πολίτες δεν θα κατανοήσουν ότι ο κόσμος μεταβάλλεται ταχύτατα και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εντάξουμε όλοι μας ε, τη γνώση και να την επικεντρώσουμε στα προβλήματα αυτά. Τέλος. Ακούσαμε πολλά για τις συνέργειες και θέλω να επισημάνω κάτι. Να υπενθυμίσω ότι ο απόλυτος στόχος του ΙΣΕΦ είναι μειώσουμε το κενό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, των 30. Να μειώσουμε λοιπόν τις διαφορές αυτές. Ο ρόλος του Horizon είναι η αριστεία. Αλλά πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλο δυναμικό για να βρούμε τρόπους ε, για το πώς θα συνενωθούν αυτοί οι στόχοι. Το θέμα δεν είναι μόνο ορίζοντας. Το θέμα είναι το πώς μπορούμε να βρούμε και στα αγροτικά ταμεία τους τρόπους να προωθήσουμε τους ίδιους στόχους. Τέλος, να πω δεν λόγια προς την Επιτροπή. Είναι σημαντικό αυτά που ακούσαμε και όχι μόνο το πώς τα είπε, αλλά και πού τα είπε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ στο Κατοβίτσο για την τεχνολογία που επικεντρώθηκε στην καινοτομία, όπου ξεκίνησε λέγοντας και παραθέτω ότι η θεμελιώδης επιστήμη θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα του μέλλοντος της Ευρώπης τέλος της παράθεσης. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει απόλυτα το τι, το τι γίνεται. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ θεμελιώδους και εφαρμοσμένης επιστήμης. Χρειάζεται σωστή ισορροπία. Γιατί ο Επιτροπός είπε πραγματικά ότι δεν γνωρίζουμε τι μας ξημερώνει αύριο ποια θα είναι το επόμενο μεγάλο θέμα. Γι' αυτό το Horizon Europe θα πρέπει να το διαχειρίσουν οι επιστήμονες. Το υποστηρίζω αυτό απόλυτα και στα σχόλιά μου ανέφερα διάφορους τομείς. Τους τομείς εκείνους όπου πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ υποστήριξη στις τρέχουσες προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω να δώσω το λόγο στον Διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής και Συντονισμού, τον κύριο Φαντενμπέργκε, να κάνει τα καταληκτικά του σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σπάνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει τον τελευταίο λόγο στο Κοινοβούλιο. Πραγματικά νιώθω πολύ προνομιούχος που μου συμβαίνει. Ε, κυρίες και κύριοι ε, ευρωβουλευτές, ε, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα ότι το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη είναι ένα μεγάλο, μικρό πρόγραμμα. Φαίνεται μεγάλο στον προϋπολογισμό, αλλά είναι μάλλον μικρό και νομίζω ότι ο Ντομινίκ Γκελέκ το τεκμηρίωσε αυτό σαφέστατα. Υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες για πάρα πολύ κόσμο, για πολλούς φορείς σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει αυτό το πρόγραμμα και βεβαίως δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα όλου του κόσμου, όσο μεγάλο είναι και να είναι ένα πρόγραμμα. Ε, εμείς αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε, που θέλαμε να προωθήσουμε όταν σχεδιάσαμε το πρόγραμμα αυτό είναι μια μεγιστοποίηση του αντικτύπου αυτού του προγράμματος για την οικονομία και για την κοινωνία. Ε, ε, δηλαδή θέλουμε κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των επενδύσεων που μπορούμε να επιτύχουμε μέσω του προγράμματος Horizon Ευρώπη. Το θέμα είναι τι αντίκτυπο θέλουμε να επιτύχουμε, τι αξία θέλουμε να ε, υπάρξει για την κοινωνία και την οικονομία και όχι ποιο θα πάρει περισσότερα, ε, ποιοι τομεί θα πάρουν περισσότερα, περισσότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιο πολλά οι μεγάλες επιχειρήσεις, ε, είναι αυτό έναντι εκείνου και σε ποιο σημείο της Ευρώπης. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ ήθελα να συνεχίσω αυτό που είπε ο Ντομινίκ Γκελέκ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουμε λίγο περισσότερο σαν τους Κινέζους, να είμαστε λίγο πιο... να χρησιμοποιούμε λίγο περισσότερο τη στρατηγική. Ε, δηλαδή, να μην δίνουμε έτσι απλόχερα τα χρήματά μας, να υπάρχει τέλος πάντων μια κατεύθυνση για το τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό ε, το ε, πρόγραμμα που είναι τόσο ουσιαστικό για το μέλλον της Ευρώπης. Περνάμε λοιπόν από ένα πρόγραμμα ε, βασικό σε ένα πρόγραμμα επενδυτικό για να δείξουμε ακριβώς πώς μπορεί να υπάρχει αντίκτυπος για την κοινωνία, για τους πολίτες και για την οικονομία. Και συμφωνώ απολύτως ε, με την κυρία Βίρινγκ ότι ο αντίκτυπος για τους πολίτες είναι μεγαλύτερος από αυτό που θα μπορούσε να ε, πάρει ο πολίτης ξεχωριστά μεμονωμένα από κάθε πρόγραμμα. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να υπάρχει, να επιτύχουμε τους στόχους ε, αηφόρου ανάπτυξης. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ανταγωνιστικότητά μας στην Ευρώπη, για την Ευρώπη, να υπάρχει μεν, αλλά να συνάδει αυτό με την αηφόρου ανάπτυξη ε, παγκοσμίω. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε μια συστημική προσέγγιση. Δεν ε, σκεφτόμαστε με τη λογική των τομέων ή τομέων του επιστητού, γιατί αυτό μπορεί να αποξενώνει κάποιες ερευνητικές κοινότητες ή κάποιους ε, τομείς οι οποίοι δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσουν το πού ακριβώς βρίσκονται σε αυτό το πρόγραμμα. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα, να συμπεριλάβουμε περισσότερους ε, ε, τομείς και να υπάρχει μια συνδημιουργία των λύσεων για το μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς προτείναμε την ιδέα, την έννοια των αποστολών, να μην είμαστε εμείς που είμαστε στις Βρυξέλλες αυτοί που θα καθορίζουμε αυτές τις αποστολές αλλά να δούμε, το, να δούμε περιοχές της Ευρώπης, στις οποίες θα μπορούσαν να υπάρχουν αυτές οι αποστολές και τότε εκεί επιτόπου αποκινούμε που τους πολίτες να σχεδιαστούν ε, οι ε, αποστολές αυτές για να επιτευχθεί και ο στόχος. Αυτό που επίσης θέλουμε να κάνουμε είναι να συμπεριλάβουμε τους πολίτες στην επιστήμη και στην έρευνα. Ε, τα, τους τελευταίους μήνες Είδαμε στη Φλάνδρα εδώ στο Βέλγιο ένα καταπληκτικό παράδειγμα. 20.000 οικογένειες συμμετείχαν σε μια επιστημονική προσπάθεια του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας ε, για ε, να μετρηθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. 20.000 ε, οικογένειες ε, συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο στη συνέχεια προβλήθηκε πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό και για την κοινωνία και για τους πολίτες και για την επιστήμη και την έρευνα. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω μια έκκληση. Μην κάνουμε αντιπαράθεση τεχνολογία εναντί μη τεχνολογίας. Ε, όλες τις μορφές καινοτομίας τις χρειαζόμαστε και αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε με αυτό το πρόγραμμα είναι να αρχίσουμε να αλλάξουμε κάπως την καινοτομία, ε, να την μεταμορφώσουμε κάπως. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που επιφέρει την αλλαγή που θέλουμε να επιτύχουμε. Ένα συνδυασμό πολλών προγραμμάτων και πολλών τομέων ε, ε, οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Ε, είναι μόνο με τη συνεργασία αυτή που μπορούμε να επιτύχουμε σε αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα. Χρειαζόμαστε συνεπείς προσπάθειες με όλα τα προγράμματα Παράλληλα, γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να βλέπουμε μεμονωμένα κάθε τεχνολογία ή κάθε τομέα, ε, κάθε τομέα μεμονωμένα. Ε, πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Γι' αυτό ε, πιστεύω ότι η τεχνολογική η ηγεσία και συμφωνώ απολύτως με την κυρία Χελίτσκα είναι αυτή που θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης στο μέλλον. Δεν είναι μιλώντας ε, για την τεχνολογία που θα κερδίσουμε, ε, με την επένδυση θα κερδίσουμε για να εξασφαλίσουμε ότι και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Οι υπόλοιποι να ακολουθούν εμάς. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν ε, λίγο κοντόφθαλμο να πούμε ότι παραγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επένδυση ε, σε ε, επιστημονική ηγεσία. Εμείς θέλουμε, θέλαμε να αυξήσουμε το ERC που είναι αυτό που έχει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό στο πρόγραμμα και θα θέλαμε σε γενικές γραμμές να μην δούμε αντιπαράθεση μεταξύ ε, της θεμελιώδους και της εφαρμοσμένη έρευνα. Ξέρω ότι είναι εύκολο να μιλάμε με αυτού τους όρους, αλλά ούτω ή άλλω από τον ορίζοντα 2020 δεν υπάρχει αυτή η διάκριση. Δεν θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη αυτή η ορολογία πρέπει να σκεφτόμαστε ποιο θέτει το θεματολόγιο. Είναι η επιστήμη, είναι η κοινωνία ή είναι η καινοτομία. Και δεν έχει σημασία αν είναι βασική εφαρμοσμένη. Χρειαζόμαστε όλη αυτή την έρευνα. Και κάποια λίγα στοιχεία επιτρέψτε μου επιπλέον και μετά θα κλείσω, Πρόεδρε. Φυσικά, το να μοιραζόμαστε την ε, αριστεία και η πιο ευρεία συμμετοχή είναι κάτι που προφανώς μας απασχολεί. Νομίζω ότι αποτελεί μια πρόκληση και μια ανάγκη με την οποία όλοι θα πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε το μερίδιο αυτό. Να μοιραζόμαστε πιο πολύ την αριστεία, όπως το ονομάζουμε στο Horizon Europe. Θέλουμε λοιπόν να ανοίξουμε πιο πολύ αυτή την πρόεδρο, να ε, εκφράσουμε εκ νέου τις προκλήσεις της κοινωνίας ε, για να δοθεί νέα πνοή και νέες πρακτικές ε, ε, στο πρόγραμμα, να εργαστούμε πιο πολύ σε ό,τι αφορά τη σφραγίδα αριστείας, θέλουμε να επενδύσουμε προκειμένου οι συνέργειες να διαδράσουν, να αλληλεπιδράσουν και με άλλα προγράμματα, να καταρτήσουμε κοινέ στρατηγικέ και ούτω καθεξής. Αλλά πιστεύω και υπάρχει γενική ομοφωνία ότι θα πρέπει να διατηρηθεί και η αριστεία ως βασικό κριτήριο και η βασική, ο βασικός στόχος του προγράμματος αυτός και παραπεπτόντως η αριστεία δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κανείς άριστος ή όχι. Η αριστεία στα πλαίσια του προγράμματος πλαίσιο είναι κάτι το οποίο πρέπει να πετυχάνουμε, να πετυχαίνουμε κάθε φορά, με κάθε καινούργια πρόταση και χαίρομαι κύριε Νίκα που σας αναφέρω ότι έχουμε αρνηθεί διάφορες δημοσιεύσεις, όχι μόνο με το σύστημα προ... πρώτερης αξιολόγησης, αλλά και με την κανονική αξιολόγηση. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και δεν θα αντιστάσουμε το ξανακάνουμε. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους όμως να εξασφαλίσουμε ότι τα δίκτυα αυτά τα οποία υπάρχουν είναι ανοιχτά. Και είμαστε οι πρώτοι που να ζητούμε λύσεις, χωρίς ωστόσο να διακυβεύουμε την αριστεία μας. Επίσης, είπατε, Πρόεδρε, πώς μπορούμε να είμαστε και ανοιχτοί και να διατηρήσουμε την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων στην Ευρώπη και να είμαστε να κρατήσουμε τα επίπεδο των αποτελεσμάτων μας. Ε, το κάνουμε εξασφαλίζοντας ότι σε κάθε επίπεδο, σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, βελτιώνουμε τις ε, συνθήκες πλαίσιο προκειμένου και οι επιστήμονες και οι καινοτόμοι να μπορούν να εργαστούν, να έχουν ένα δυναμικό απόδοση των επενδύσεων τους. Ε, αν το κάνουμε λοιπόν αυτό, σας ε, διαβεβαιώ ότι η Ευρώπη μπορεί να καταστεί ένα τόπος όπου ανθούν όλες αυτές οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε λοιπόν που είσαστε τόσο γενναιόδωρος στο χρόνο που μου δίνετε ο κύριος Έλερ μας ρώτησε σε, κάποιο χρονικό σημείο εξ ονόματος του κυρίου Βελίτσικα το τι κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ηγετική στον κόσμο. Τρία πράγματα, η ταχύτητα, η κλίμακα και το πεδίο εφαρμογή. Κινώντα λοιπόν το τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις, ταχύτητα, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε γρήγορη συμφωνία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχει κενό στη μετάβαση από το Horizon 2020 στο ορίζοντα Horizon Europe Scale, ε, ε, κλίμακα, προϋπολογισμός. Είναι μικρός ο προϋπολογισμός. Ακόμα και με 120 εκατομμύρια δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από το πόσο αυτό και εφαρμογή εφαρμογής, έρευνα και καινοτομία. Χρειαζόμαστε όλες ε, τις πτυχές, όλους τους τομείς. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά στην οικονομία και στην κοινωνία προκειμένου να συμβάλλουμε στην ε, επιτυχία του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, λέει και ο Πρόεδρος. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Έλε, θα θέλει να πάρει το λόγο για να κάνει τα καταλεκτικά του σχόλια. Κοιτάξτε, δεν θέλω να υπερβάλλω γιατί έχουν κουραστεί και οι Να σας καλέσω στο τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης να μας βοηθήσετε ο λόγος για τον οποίο δεν ε, μπόρεσα να παρευρεθώ εδώ το τελευταίο μισάωρο είναι ότι το Συμβούλιο δεν θα ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση των τελευταίων χρόνων. χρονικά και άρα αυτό θα περάσει στο επόμενο κοινοβούλιο. Δεν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά του χρόνου. Θα πρέπει να περιμένουμε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, της νέας ε, επιτροπής, συγγνώμη, και τελικά θα καταλήξουμε να τα κάνουμε όλα αυτά τέλη του 2020. Άρα, δεδομένων των όσων μας είπατε, ότι επίπεδο φιλοδοξίας και να έχουμε, ό,τι προτεραιότητες και να θέτουμε, ό,τι επιπρόσθετη πρόθεσε και να εκφράζουμε, όσο ευρέως και να θέλουμε να τοποθετηθούμε, αυτό που είναι σαφές στον μεταβαλλόμενο κόσμο, σε έναν κόσμο που υπάρχει ανταγωνισμό, σε έναν κόσμο που, ο κόσμος, που δεν ε, περιορίζονται οι πολίτες στη χώρα τους, στην ήπειρό τους. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι χάνουμε στον ανταγωνισμό και θα ήθελα να σας καλέσω το κοινοβούλιο αυτό τίθεται και βάση αλλαγή της νομική βάση. Η φιλοδοξία του Κοινοβουλίου είναι να συλλέξει όσο πιο πολλούς πόρους γίνεται. Το πρώτο σημείο προκειμένου να υπάρχει μια κανονική νομική διαδικασία. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι μετά το Brexit, το οποίο δεν είναι ενδεχομένως ιδανικό, το σημείο τομή είναι ότι θα επικεντρωθούν όλες στην Ευρώπη. Και αν το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια φιλόδοξη πρόταση, η οποία δεν βρίσκει αντίθετα κανένα θεσμικό όργανο. Τελικά καθυστερούμε μέχρι τέλη του 2020 την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Και άρα θα ξεκινήσει από το 2022-2023. Η αντίληψη για τον αντίκτυπο του Brexit θα είναι τεράστιος. Γιατί δεν θα είμαστε πλέον επί όρους. και το επιχείρημα ότι όταν υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας οι αποφάσεις είναι τόσο πιο γρήγορες που τελικά παρέχεται οικονομική ευημερία στο λαό θα ενισχυθεί. Θα δοχεί η εντύπωση ότι θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρο τι δημοκρατικές φιλοδοξίες. Το θέμα αυτό ξεπερνάει το θέμα του προπολογισμού, το θέμα της έρευνας. Το συγκριτικό λοιπόν μειονέκτημα μιας επαχθούς αργής διαδικασίας θα δώσει την εντύπωση σε παγκόσμιο επίπεδο ότι μένουμε πίσω. Όχι μόνο σε αριθμητικά στοιχεία, αλλά ως προς το κύρος μας, ως προς ε, τα έργα τα οποία μπορεί να πετύχει μια δημοκρατία. Άρα, έχω να απευθύνω την εξής έκκληση. Δεν πρέπει να τα δούμε όλα αυτά ξεχωριστά. Να μείνουμε σε επίπεδο μικρολόμπινγκ, μικροδιαχείρισης ε, με ιτημένους και κερδισμένους. Θα χάσουμε όλοι μαζί. πρέπει να είναι αυτή η Ευρώπη μας, η Ευρώπη που θα αυξήσει τον προϋπολογισμό, που θα δηλώνει ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν ακολουθούμε μόνο τον τεχνοκρατικό τρόπο για την ε, μεταμόρφωση των στοιχείων αυτών. Θέλουμε ένα αποτέλεσμα όχι μόνο τεχνικά άρτιο, θέλουμε ουσιαστικές αλλαγές. Νομίζω ότι αυτό που διακυβεύεται είναι ο τρόπος άσκησης πολιτικής στην Ευρώπη σε σχέση με το πώς ασκούνται η πώς ασκείται πολιτική στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι και οι δύο οι σύντες παρουσίασαν τις ιδέες τους με ευρύτερο τρόπο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω τον κύριο Φανεμπέρχε τον καθηγητή Γιάννου Μπουνίσκι από το Διεθνές Ινστιτούτο της Βαρσοβίας, την, τον κύριο Ντομινίκ Γκέλεκ, επικεφαλής ε, του ΑΣΑ για τα θέματα πολιτικής, ε, την κυρία Σαμπίνε Χερλίτσκα και τον Γιάνν Παρνόφσκι, Γενικό Γραμματέο των, ε, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Ήταν χαρά μας και τιμή μας που τα συζήτησαμε αυτά από κοινού. Εξαντλήσαμε το χρονικό μας όριο, ωστόσο ήταν τόσο ευρία η σύνθεση της ομάδας που θεωρώ ότι σίγουρα θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά και είμαι βεβαίως ότι το θέμα αυτό θα το εξετάσει με πολύ πιο σωστό τρόπο το επόμενο κοινοβούλιο. Αύριο στις 9 συντονιστές και στις 10 ψηφοφορίες. Τα λέμε αύριο.